Να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίασή μας. Έχουμε μία ώρα, ουσιαστικά μέχρι τις 10, αλλά έχουν μείνει 45 λεπτά για την πρώτη. Το πρώτο θέμα μας που είναι η ανταλλαγή απόψε, ένα θέμα πολύ σημαντικό. Να ξεκινήσουμε με την έκρηση της μερίσιας διάταξης. Σας ενημερώνω ότι ο κύριος Ρίλε, συντάκτης γνωμοδότηση για τη συμβάση παραχώρησης ε, προβλέπεται για τις 5 και μισή κύρα συγκεκριμένα δεν μπορεί να έρθει το απόγευμα, οπότε θα προσπαθήσουμε μετά την ψηφοφορία, αν τελειώσουμε νωρίτερα, να το εξετάσουμε. Αλλιώς θα πρέπει να γίνει το μεσημέρι. Τουλάχιστον έχουμε την αλλαγή απόψεων και να προτείνουμε μια προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Δεν μου έχει υποβληθεί κάποιο άλλο αίτημα ως προς ε, τροποποίηση μερισιάς διάταξη, άρα μπορούμε να την εγκρίνουμε. Θα ήθελα να σα ενημερώσω επίσης ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μα και να σας ενημερώσω πως πάντοτε κάνω στην αρχή ότι θα πρέπει να θεωρήσετε ενδεικτικά τα χρονοδιαγράμματα γιατί κάποιες φορές καθυστερούμε, κάποιες φορές πηγαίνουν λίγο πιο γρήγορα. Να είστε λοιπόν έγκαιρα εδώ για τα σημεία που σας ενδιαφέρουν. Σημείο 2 στην μέση διάταξη, έγκριση των πρακτικών. Έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά της συνεδρίασης στι 11ης-12ης η ιουλιου Θα θεωρηθούν εγκεκριμένα, εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις. Και έχουμε δυστυχώς ε, ένα πρόβλημα τα πρακτικά της 17 η 18 ης δεν είναι διαθέσιμα Σεπτεμβρίου. Ανακοινώσει πρέπει δεν έχω ανακοινώσει. Άρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Άκρος σημαντικό θέμα για την πολιτική μας. Μια ανταλλαγή απόψε με τον Κώστα Χατζηδάκη, Έλληνα Υπουργό Ανάπτυξης. Στην ελληνική κυβέρνηση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Δίνω απευθείας τώρα στον Κωστή Χατζηδάκη. Ό,τι θεωρεί ότι είναι σημαντικό να μας το μεταφέρει, παρακαλώ, Κωστή, έχεις το λόγο και μετά θα έχουμε και μια χώρο για, και χρόνο για ερωταπαντήσεις. Thank you, President. I would like to... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω oh. τις ευχαριστίες μου προς την πρώτη Ντανούτα Χούμπνερ, τους συναδέλφους, όλους παρόντες. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι νιώθω πάρα πολύ οικία εδώ. Υπήρξα μέλος του Κοινοβουλίου για 13 χρόνια, από το 1994 στο 2007. Ήμουν εισηγητής και για το προηγούμενο πακέτο για τη συνοχή, για τις ρυθμίσεις σχετικά και τους κανονισμούς σχετικά με το Ταμείο Συνοχής. Έξω και όπως σας προείπα νιώθω πάρα πολύ οικία με όλα εκτός από το κτίριο που είναι καινούριο για μένα. Δεν το έχω ξανά επισκεφθεί. Πολλά μέλη τη επιτροπή όταν και εγώ ήμουν ευρωβουλευτή, ε, βλέπω να έχουν παραμείνει. Τροπή Κωνσταντς, λέει Ντάντα Χούμπνερ. Λοιπόν, αυτό που έχει αλλάξει δυστυχώ, Άρδιν, είναι η όλη οικονομική κατάσταση. Το 2007, όταν έφυγα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη δραματική αυτή κρίση. Ασφαλώς αυτό ισχύει για τη χώρα μου, διότι είμαστε εν μέσω αυτής της πάρα πολύ βαριάς κρίσης και πρέπει να αγωνιστούμε για να την ξεπεράσουμε το συντομότερο δυνατόν. Και θα ήθελα να ξεκινήσω τη σύντομη ομιλία μου, αναφέροντας τα εμπόδια με τα οποία έρχομαστε αντιμετώπιση στην Ελλάδα. Κυρίως αυτό που πρέπει να ξεπεράσουμε είναι εμπόδια τριών διαφορετικών μορφών. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία της χώρας. Δεύτερον, πρέπει να προχωρήσουμε με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και τρίτον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της ρευστότητα που απειλεί την οικονομία μας. Ξεκινήσω με το πρώτο ζήτημα. Το πρόβλημα εμπιστοσύνης, το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας των προσπαθειών μας. Πρέπει να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργό και τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, αλλά και ο ελληνικός λαός, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να δώσουν τον αγώνα αυτό που είναι ο αγώνας της γενιάς μας. Ξέρετε, γνωρίζουμε όλοι μας πόση μεγάλη σημασία έχει η αξιοπιστία και πρέπει να εκπλήξουμε θετικά τον κόσμο. Πρέπει να υπογραμμίσουμε την αποφασιστικότητά μας. Είναι η λέξη κλειδί, η λέξη αποφασιστικότητα για μας. Εξώ και η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να παραγνωρίσει το πολιτικό κόστος και να εγκρίνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να πείσει ότι δεν είμαστε χαμένη υπόθεση, ότι είμαστε εδώ θα συνεχίσουμε να είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης, διότι είμαστε Ευρωπαίοι και θα παραμείνουμε στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Και αν συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε την ίδια αποφασιστικότητα, θα έχουμε ήδη ε, πετύχει κατά 50%. Εγώ νομίζω ότι μετά τις εκλογές έχει αλλάξει το κλίμα. Είμαστε αποφασισμένοι λοιπόν να πολεμήσουμε κάθε μέρα για να αναστρέψουμε πλήρως το κλίμα. Το πρώτο εμπόδιο λοιπόν, πρώτος πυλώνας της όλης προσπάθειας είναι ο αγώνας για την ανάκτηση της χαμένης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν προκειμένου να πετύχουμε και παραλαμβάνουμε να εκπλήξουμε θετικά τις αγορές, τους επενδυτές και τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Έπειτα, έχουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Άκρο σημαντικό ζήτημα. Πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών. Η φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε το Υπουργείο των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Ανακοινώσαμε τον Αύγουστο 10 συγκεκριμένους στόχους για διάφορα ζητήματα που πηγαίνουν από τις ε, ιδιωτικοποιήσεις μέχρι τους, δημόσιους, τους διαγωνισμούς, της δημόσιες απελευθέρωση αγορών μέχρι διαχείριση διαρθωτικών ταμείων. Όλοι αυτοί οι στόχοι έγιναν δεκτοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα την ίδια ημέρα. Αποφασίσαμε να ορίσουμε διευθυντές έργων, συντονιστές για τον κάθε στόχο. Έχουμε επίσης καθορίσει σαφή χρονοδιαγράμματα προκειμένου να εκπληρώσουμε τους στόχους και να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Και ακόμη είμαστε μέσα στις προθεσμίες. Αυτό το αναγνωρίζει η Τρόικα. Μπορώ να σας πω, ως παράδειγμα, ορισμένα πράγματα. Πρώτον, νέος επαναπτικός νόμος καταθέσαμε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για να βελτιωθούν ταχείες διαδικασίες, fast track. Έχουμε οργανώσει το Υπουργείο ώστε να εγκρίνει τις στρατηγικές επενδύσεις ως μία νέα αρχή αδειοδότησης. Προχωρήσαμε επίσης δίνοντας στους επενδυτές τη δυνατότητα της αυτοαξιολόγησης για να περιοριστεί η γραφειοκρατία, για να γίνει η χώρα μας φιλική προς τις επενδύσεις. Επίσης υπογράψαμε μία σύμβαση με τον ΩΣΑ, ώστε να μπορούμε την εργαλειοθήκη για την αξιολόγηση ε, να την ε, να, το, να την αξιοποιήσουμε και να μην έχουμε πλέον εμπόδια. Θα μας βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή ο Διεθνής Οργανισμός γιατί γνωρίζουμε ότι η απελευθέρωση της οικονομίας μας είναι κάτι παραπάνω από σημαντική και για την ανταγωνιστικότητα της χώρας, αλλά και για τους καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά τις ε, προμήθειες, προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά, να ε, πληρώσουμε αυτό το χάσμα με κάποια μέτρα ηλεκτρονικών προμηθειών ή procurement και προχωρούμε και με τις ιδιωτικοποιήσεις. Ε, για παράδειγμα, έχουμε τους σιδηροδρόμους στο Υπουργείο μας και διαπραγματευόμαστε με την Κομισιόν για να λύσουμε το πρόβλημα των κρατικών ενισχύσεων. Έτσι θα μπορέσουμε, εν συνεχεία, να συνεχίσουμε τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων. Εδώ σταματώ με τα παραδείγματα, είναι άριθμοι και σε πολλά μέτωπα τα παραδείγματα που θα μπορούσα να σας δώσω, αλλά σας είπα ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και καταλαβαίνουμε ότι αφού αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία της χώρας, έχει εξαιρετική σημασία να προχωρήσουμε με τις διαρθρωτικές αυτές μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα βοηθήσει τη χώρα να ξεπεράσει όλα αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα. Αμφότερες προσπάθειες αυτές δηλαδή, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και διενέργεια των απαραίτητων διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων εξαρτώνται από εμά στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Υπάρχει και ένα τρίτο εμπόδιο, όμως, το οποίο δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται, θα έλεγα, κατά βάση από εσάς, από τις Βρυξέλλες. Εννοώ τη ρευστότητα. κατά πάσα πιθανότητα είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μετά το κούρεμα της προηγούμενης άνοιξης, το τραπεζικό μας σύστημα είναι ένα άδειο ταμείο θα έλεγα πλέον, ένα κενό κέλυφος. Δεν λειτουργεί. Γι' αυτό η συμφωνία με την Τρόικα προκειμένου να πετύχουμε την επανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού μας τομέα είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ρευστότητα. Έχουμε όμως και τα καθυστερούμενα, τα χρήματα δηλαδή που πρέπει να καταβάλουμε στον ιδιωτικό τομέα. Και νομίζω ότι το στόχο αυτό μπορούμε να τον πετύχουμε πάλι βασιζόμενοι στην τρόικα, εξαρτώμενοι από την τρόικα. Χωρίς ρευστότητα δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις προσπάθειές μας. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη της οικονομίας μας. Και δεν πρέπει να τρέχουμε αυταπάτες. Τα μέτρα λιτότητας πρέπει να συνδυαστούν με μέτρα για την ανάπτυξη, αναπτυξιακά μέτρα. Αλλιώς τα μέτρα λιτότητας δεν θα αποδώσουν. Όπως σας είπα, είμαστε έτοιμοι τα σκληρά αυτά μέτρα λιτότητα να τα υιοθετήσουμε. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι χωρίς ένα πραγματικό αναπτυξιακό πακέτο για τη χώρα μας δεν θα αποδώσουν τα μέτρα, δεν θα λειτουργήσουν. Και η αποτυχία της Ελλάδας θα είναι αποτυχία της Ευρώπης και δεν μπορεί αυτό να αποτελεί επιλογή. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη συμφωνία με την Τρόικα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ρευστότητα. Και έτσι να μπορέσει να επανεκκινήσει ο τραπεζικός μας τομέας. Ταυτόχρονα δε η Ευρώπη πρέπει και αυτή να τιμήσει τις υποσχέσεις της για το λεγόμενο σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα. Δεν μιλάμε για φρέσκο χρήμα από άλλες ε, κεφαλαιοαγορές. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τις ναι. δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας από τα άλλα εθνικά κοινοβούλια για να εγκρίνουν ε, την χορήγηση ενισχύσεων προς την Ελλάδα, αλλά εδώ μιλάμε για μια πραγματική ευρωπαϊκή προσέγγιση από τις Βρυξέλλες. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γνωρίζω ότι έχετε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, για να τα πω έτσι ευγενικά τα πράγματα για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Πρατισλάβα για να συζητήσω το ζήτημα αυτό με τους φίλους μας, τους φίλους της συνοχής, όπως τους λέμε. Αγαπητοί φίλοι, αυτό που θα συμβεί με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και την Ελλάδα θα έλεγα μάλλον αυτό που γίνεται είναι κάπως περίεργο. Δηλαδή είμαστε η χώρα με την πλέον δραματική μείωση τουλάχιστον σε σχέση με την περσίνη πρόταση κομισιών. έχουμε μία μείωση της τάξης του 40% σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Φαντάζομαι κατανοείται πλήρως ότι δεν μπορούμε την προσέγγιση αυτή να την δικαιολογήσουμε. Καταλαβαίνω ότι η Κομισιόν εφαρμόζει τη μεθοδολογία του Βερολίνου, η οποία υιοθετήθηκε το 1999 και λαμβάνει στοιχεία, υπόψη τη στατιστικά στοιχεία από το 7 στο 9, πριν την κρίση δηλαδή. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία όμως δεν έχουν καμία σχέση πλέον ε, με την ελληνική πραγματικότητα. Γνωρίζετε ότι φέτος είναι το πέμπτο συναπτό έτος ύφεσης η οποία κινείται στο 27%. Σορευτικά. Αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Όταν λοιπόν τον επόμενο μήνα αποφασιστεί η κατανομή των κονδυλίων και δεν λαμβάνεται υπόψη αυτός ο πολύ σημαντικός παράγοντας καθόλου, πώς θα γίνει. Πρέπει να παρουσιάσουμε στους πατριώτες μας στην Ελλάδα ότι η Ευρώπη έδειξε την αλληλεγγύη της. Μείωσε κατά 40% το πακέτο. Μιλάμε για δραματική μείωση, κάθετη, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ήρθα εδώ λοιπόν για να σας πω ότι ναι, είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε για τη χώρα μας. Γιατί είναι παραλαμβάνω ο αγώνα που δίνει η γενιά μα, ο αγώνα μια γενιά ολόκληρη. Είμαστε εδώ αποφασισμένοι και ο Πρωθυπουργό προσωπικά να αγνοήσουμε το πολιτικό κόστο και να υιοθετήσουμε όλα τα απαιτούμενα φορολογικά μέτρα για την αντιμετώπιση τη κρίση. Ναι, είμαι εδώ για να σα πω ότι λάβαμε την απόφαση να προχωρήσουμε με όλες τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για να απελευθερώσουμε την οικονομία μας και να κάνουμε την Ελλάδα ανταγωνιστική. Ναι, είμαστε αποφασισμένοι να επομιστούμε το πολιτικό κόστος και να προχωρήσουμε. Ταυτόχρονα όμως χρειαζόμαστε και τη δική σας αλληλεγγύη. Η λιτότητα πρέπει να συνδυαστεί με μια αναπτυξιακή δέσμη μέτρων, πραγματικών αναπτυξιακών μέτρων. Προκειμένου να το πετύχουμε, το στόχο αυτό, ίσως το πρώτο πράγμα που πρέπει μαζί να κάνουμε είναι να έχουμε ένα πραγματικό πακέτο συνοχής για την Ελλάδα για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Ουσιαστικά αυτά είναι όσα είχα να σας πω. Δεν θέλω να επεκταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες. Η Ελλάδα χρειάζεται την αλληλεγγύη της Ευρώπης. Αυτό είναι βέβαιο. Είμαι βέβαιος ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κατανοητό το μήνυμα αυτό. Ξεκάθαρα και περίφαστα λοιπόν σας λέγω ότι είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τη δουλειά που μας αναλογεί. Θα το δείτε. Θα δείτε πόσο αποφασισμένη είναι η ελληνική κυβέρνηση τους προσεχείς μήνες. Έχουμε διδαχθεί από το παρελθόν έχουμε αποφασίσει να γίνουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα, μια ανταγωνιστική οικονομία. Αποφασίσαμε να γνωρίσουμε επαναλαμβάνω, το πολιτικό κόστος, ωστόσο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μόνοι μας. Η Ελλάδα χρειάζεται την αλληλεγγύη της Ευρώπης. Είμαι βέβαιος ότι αυτή την αλληλεγγύη θα μας την προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας και θα ήθελα όποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο να μας κάνει ένα νεύμα. Βλέπω ότι έχουμε εδώ και πολλούς συναδέλφους από την Ελλάδα Θέλω να σας πω το εξή ότι αν έχετε καλοσύνη μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά στην ερώτησή σας, γιατί μετά ο, ο κ. Χατζηδάκης δεν θα έχει χρόνο να απαντήσει. Πραγματικά έχουμε μόνο μία ώρα στη διάθεσή μας. Γι' αυτό μην κάνετε ερω... μεγάλες ομιλίες, απλά να υποβάλλετε ερωτήσεις. Ε, Λαμπέρ, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι μπορώ να βαδίσω στα βήματα που μου έμαθε ο Κώστας, ε, εγώ το έχω μάθει τουλάχιστον. Ε, θα είμαι σύντομος. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ. Υπάρχουν κάποια μυστικά και κάποια πράγματα που έχουν αλλάξει από την τελευταία περίοδο. Τώρα υπάρχει δυνατότητα συναπόφασης με το Συμβούλιο και θέλω να πω το εξής, ότι όταν ήσουν εσύ εδώ υπήρχε ίσως η ίδια διαδικασία, αλλά απλά άλλαξα κάποια πράγματα και ακόμα εξακολουθεί να είναι μυστικό το πώς το κατάφερες αυτό, ε, γιατί δεν είναι εύκολο να αγωνιστεί κανείς με το Συμβούλιο. Πάντως έχουμε κάνει εντωμεταξύ αυτή την εμπειρία. Είναι σημαντικό να μας δώσεις ε, άμεσες πληροφορίες. Επειδή θέλω να είμαι σύντομος, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώς αισθάνεσαι οι αλλαγές οι οποίες πρόσφατα έγιναν στους κανονισμούς. Οι αλλαγές αυτές έγιναν για να μπορεί η Ελλάδα να απορροφήσει τα κονδύλια που προβλέπονται ειδικά για αυτήν. Είχαμε εδώ διάφορες συναντήσεις με την Task Force. Πριν από 1,5 χρόνο πήγαμε στην Ελλάδα για να δούμε πώς λειτουργεί η κατάσταση. Ίσως λοιπόν μπορείς να μας δώσεις ε, μια εικόνα, να μας ενημερώσεις για τα θέματα της περιφερειακής πολιτικής. Και τελευταία μου παρατήρηση σχετικά με την αλληλεγγύη. Πράγματι, ε, είναι απόλυτα σωστό αυτό που είπες. Εδώ έχεις τους φίλους της ε, συνοχής, τους οπαδούς μιας ε, κοινής ε, φιλελεύθερης πολιτικής ε, σε θέματα συνοχής. Έχουμε λοιπόν την εξής κατάσταση. Έχουμε κοινούς στην Ευρωζώνη οι οποίοι ασχολούνται με τα οικονομικά προβλήματα αυτή τη στιγμή και φτάνουν μάλιστα να λένε ότι μέσα στην ίδια την Ευρωζώνη θα πρέπει να επηρεάσουμε καλύτερα θέματα προπολογισμού. Αυτό όμως θα είναι το τέλος της ε, πολιτικής ε, συνοχής. Εδώ υπάρχει μια κοινή προσέγγιση. Δουλεύουμε στο πνεύμα που παρουσίασες και εσύ και δεν θα υποχωρήσουμε. Η Κωνσταντσε. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είναι χαρά που σας βλέπω και πάλι εδώ και σας εύχομαι πραγματικά επιτυχία ε, προσωπική για τη δουλειά σας, για τη χώρα σας και μπορείτε να είστε σίγουρος ότι η Περιφερειακή Επιτροπή θα στηρίξει την Ελλάδα στο μέλλον. Όπως είπε ήδη ο Λάμπερτ, σας ε, παρακολουθούμε και σας παρακολουθήσαμε τότε ε, σε αυτά που κάνετε για το γενικό κανονισμό. Ε, τώρα έχουμε την συναπόφαση. Τα πράγματα ίσως να μην είναι πιο εύκολα, πάντως προσπαθούμε και σίγουρα πρέπει να προσπαθήσουμε για το δημοσιονομικό πλαίσιο και τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Όμως το Συμβούλιο ε, προσπαθεί να περικόψει τα κονδύλια για τη σύνοχη. Αυτό είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε και τώρα και η Γερμανίδα Καγκελάριος έχει μάθει ότι δεν μπορεί να υπάρχει μόνο λιτότητα αλλά χρειάζεται και ανάπτυξη και η ανάπτυξη προκύπτει μέσα από τη συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω μία ερώτηση. Έχουμε συναντηθεί αρκετέ φορέ με τον κύριο Ράιχεμπαχ, τον επικεφαλή τη Task Force στην Ελλάδα. Μήπω μπορείτε να μα πείτε λιγάκι πώ ακριβώ ξεκίνησε η δουλειά, πώ προχωράει. Υπάρχουν δηλαδή ελπίδε που να εκφράζει η ίδια η Task Force για την Ελλάδα για την ανεργία. Τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να σας στηρίξουμε ε, στην προσπάθειά σας αντιμετώπισης της κρίσης. Ο κύριο Βλάσακ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να σε καλωσορίσω Κώστα εδώ ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ερώτησή μου είναι πολύ σύντομη. Γνωρίζω ότι έχεις πολύ στενές επαφές με την Κύπρο. Υπάρχουν κάποιες ε, ειδικέ διαπραγματεύσεις που να μπορούν να σε βοηθήσουν να λύσεις, να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Χρυσόγελος από τους Πράσινους. Προφανώ ε, έρχεσαι στο Κοινοβούλιο σε μια περίοδο που είναι πολύ δύσκολη και για την Ελλάδα σαν χώρα αλλά και για την κοινωνία και ειδικά μεγάλα κομμάτια τη κοινωνία. Και είναι όλο και περισσότερο σαφέ και στο Κοινοβούλιο το έχουμε πει πολλέ φορέ, ότι η λιτότητα δεν ανοίγει τον δρόμο για τη λύση των προβλημάτων στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε του Νότου. Πρέπει να είναι δίκαια τα μέτρα και να ε, συνδυάζονται και με μέτρα για την οικονομική αναζωογόνηση, τη μεταρρύθμιση οικονομία και την απασχόληση. Θα ήθελα να, πω, να ρωτήσω και να πω τέσσερα θέματα όμως. Ε, και εδώ η ομάδα μας έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι οι όροι του μνημονίου πρέπει να προσαρμοστούν σε ευρωπαϊκές πολιτικές και αξίες. Πολλά από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με ευρωπαϊκές οπτικές, είτε αυτό αφορά την, ε, το κατώτατο μισθό που συμφωνείται μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, είτε αφορά θέματα περιβαλλοντικά, είτε θέματα κοινωνικής συνοχής. Και αυτό δεν βλέπω ούτε σαν κυβέρνηση να το θέτεται, παρόλο ότι πολλές, πολλοί ευρωβουλευτές το θέτουν. Το δεύτερο είναι ότι ε, φοβάμαι ότι για την διέξοδο από την κρίση επιλέγονται πολιτικές που επιστρέφουν σε μια άλλη αντίληψη για το περιβάλλον. Δηλαδή και το fast track πολλές φορές πάει να παρακάμψει περιβαλλοντική νομοθεσία και αυτό είναι μια πιστοχώρηση γιατί η, η αντίληψή μας στο Κοινοβούλιο είναι ότι η κρίση αντιμετωπίζεται με σωστότερη προστασία του περιβάλλοντος και με κοινωνική συνοχή, όχι με απορρίθμιση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής. Το τρίτο που έχω θέσει και με ερώτηση εδώ είναι ότι η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ ΕΕ, και της ΕΙΑΘ, ΕΕ, όσοι δεν ξέρουν οι εταιρείε διαχείριση του νερού, που πιέζει η Τρόικα για να γίνει, αντίκειται στην, ε, στο άρθρο 258 της ε, Σύμβασης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να είναι ουδέτερη στα θέματα ε, διαχείριση του νερού από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και όρο στο μνημόνιο, αλλά και, και εσείς το είπατε πριν, για ιδιωτικοποίηση του νερού. Ενώ υπάρχει και η έκθεση του Κοινοβουλίου πρόσφατα, που βάζει ερωτήματα σχέση με αυτήν την... Ε, και τελευταίο που θέλω να μιλήσω είναι για το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μιλήσαμε, μιλήσατε πολύ για την επόμενη περίοδο, αλλά και τώρα χρήματα από το ΕΣΠΑ ή γενικότερα χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν φτάνουν εύκολα. Και ξέρουμε ότι ακόμα και εκείνες που κάνουν αίτηση στις τράπεζες για να πάρουν χρήματα, για να αναζωογονηθεί η οικονομία, δεν μπορούν να πάρουν και δεν ξέρω αν έχετε κάνει και στο επίπεδο τη χώρα αλλά και στο επίπεδο των διαβούλευση με την Κομισιόν, ορισμένε ενέργειε να φτάνουν χρήματα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είναι ο κορμό τη οικονομία, πραγματική οικονομία. Και τέλο, ε, μια, ιεράρχηση, ναι, μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων στις επενδύσεις δημόσιο-ιδιωτικές ώστε να δημιουργούν και θέσει εργασία, να μην πάνε τα χρήματα, οι δημόσιοι πόροι, μόνο σε έργα τα οποία δεν δημιουργούν προσθέμενη αξία για του ε, που είναι σήμερα άνεργοι και είναι το 25% και 55% των νέων. Ευχαριστώ. Uh, Επιτρέψτε μου να επαναλάβω αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ε, σας παρακαλώ να είστε σύντομοι η κυρία Κράτσα και μετά ο κύριος Χατζηδάκης και άλλοι τέσσερις θα λάβουν το λόγο. Καρά σας υποδεχόμαστε στην Επιτροπή μας σήμερα, ένα χώρο που το γνωρίζετε πολύ καλά και έχετε και εσείς συμβάλει σε πολιτικές που έχουν χαρακτηρίσει του Κοινοβουλίου τη δέσμευση στη συνοχή. Αναφερθήκατε πολύ σωστά στην ανάγκη για ένα πακέτο αναπτυξιακό για τη χώρα μας, το οποίο θα συνοδεύει όλες τις προσπάθειές της για δημοσιονομική προσαρμογή και για τις βάσεις μέσω μεταρρυθμίσεων για μια οικονομία πιο παραγωγική και ανταγωνιστική. Ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα από ό,τι γνωρίζω η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων της τρέχουσας περίοδου είναι σε ένα καλό επίπεδο. Θα ήθελα να μας το επιβεβαιώσετε αν είναι σωστό. Και δεύτερον, τι προβλέπετε ούτω ώστε να επιταχυνθεί η απορρόφηση που θα είναι μια τόνωση για την οικονομία οπωσδήποτε. Δεύτερον, εμείς ξέρετε έχουμε συμβάλει θετικά στην δημιουργία του μηχανισμού επιμερισμού κινδύνου που θα έδινε την ευκαιρία στην αξιοποίηση σε πόρων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη δυνατότητα μόχλευσης. Ε, έχουμε θέσει το θέμα της καθυστέρησης ε, στην Επιτροπή μας εδώ και μαζί και παρουσία του ο επικεφαλής της Task Force. Ήθελα να σας ρωτήσω πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση και σε τι μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε, γιατί θέλουμε, κύριε Υπουργέ, οι πολιτικές οι οποίες και εμείς ε, προγραμματίζουμε εδώ και προδιαγράφουμε να αποδίδουν και να εφαρμόζονται σε επίπεδο τοπικό, πόσο μάλλον στην Ελλάδα που είναι μια χώρα μέσω ανάγκης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, αν έχετε καλοσύνη γύρω στα πέντε λεπτά, δεν μπορώ να σας δώσω παραπάνω για να απαντήσετε. Κοιτάξτε, όσον αφορά στα ερωτήματα σχετικά με την διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων ε, και το ποσοστό απορρόφησης, η ερώτηση δηλαδή, της κυρίας Ζακράτσα και του κυρίου Ρόι ε, που ετέθη εκεί το θέμα αυτό. Καταρχήν να πω το εξή. Ε, υπάρχει η απλούστευση των διαδικασιών. Συμπτωματικά τελείως αύριο σε μία ε, ε, συνέντευξη τύπου θα ανακοινώσω τα βήματα που έχουμε κάνει για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να διευκολύνουμε την απορρόφηση κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Και θα συνεχίσουμε αυτές μας τις προσπάθειες. Υπάρχει μια συμφωνία που προβλέπεται στο μνημόνιο ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε ε, απλουστεύσει ολοκληρωτικά σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες. Κατόπιν, όσον αφορά, υπάρχουν και κάποια μάλλον ε, προγράμματα προτεραιότητας, ε, υπάρχουν κάποιοι διαχειριστές που έχουν επιληφθεί ειδικών προγραμμάτων προβληματικών και νομίζω ότι εκεί έχουμε σημειώσει πρόοδο και θα σημειώσουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο στο μέλλον. Τρίτον, όσον αφορά τα ποσοστά απορρόφησης κοντιλίων, το ρυθμό τους περισσότερο. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πρέπει να σας πω ότι παρά την αρνητική εικόνα που εκπέμπει η χώρα και όσον αφορά στο ρυθμό απορρόφησης κονδυλίων, είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Ε, είμαστε πάνω από το μέσο όρο απορρόφησης κονδυλίων. Δηλαδή, Είμαστε στο 45% και ο μέσος όρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο 41%. Ειδικά όσον αφορά το γεωργικό ταμείο, η απορρόφηση στην Ελλάδα είναι 49% σε σχέση με το 48% στην Γερμανία ε, και 41% που είναι ο μέσος όρος. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά στο, σε αυτό που είπε η κυρία Κρέλ στην ε, καλύτερη ε, χρήση των κονδυλίων. Η καλύτερες, ε, καλύτερη χρήση των κονδυλίων δεν σημαίνει και περισσότερη. Και συζήτησα με τον κύριο Πίτσιν και είπαμε ότι λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το κοινοτικό ΑΕΠ μειώνεται, μειώνοντας το πακέτο συνοχής, καταλήγουμε τελικά σε διπλή μείωση. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Πράγματι, συνεργαζόμαστε με την Task Force στην Ελλάδα. Η συνεργασία είναι χρήσιμη για μας. Δεν παρεμβαίνουν παντού, παρά μόνο σε ορισμένους ε, τομείς όπου η παρέμβασή τους ε, ε, προσφέρει προσθέμενη αξία. Παραδείγματος χάνει στο κτηματολόγιο ε, ή στην προαγωγή των εξαγωγών ή στην παροχή τεχνικής βοήθειας έτσι ώστε ε, να ε, απλουσευτούν οι διαδικασίες για το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Είμαστε ευτυχείς για την την εντύπωση που υπάρχει, τουλάχιστον ο κύριος Ράχεμπαχ, αυτό λέει επίσημα. Και όσον αφορά, κύριε Βλάζακ, το θέμα της Κύπρου, Ναι, η Κύπρος έχει την Προεδρία, αλλά η στενική ανάλυση ε, δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα. Ε, πρέπει να καταλήξουμε όλοι σε συμφωνία. Πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκός συμβεσμός, αλλά πραγματικά ευρωπαϊκός. Όχι συμβιβασμός ο οποίος ε, θα λαμβάνει υπόψη του εθνικιστικές απόψεις οι οποίες αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μία αμυγός ευρωπαϊκή προοπτική. Γι' αυτήν μιλάμε. Όσον αφορά στα θέματα που έδειξε ο κύριος ε, Χρυσόγελος, κοιτάξτε κύριε Χρυσόγελε, να είστε σίγουρος ότι θα λάβουμε υπόψη μας την ε, περιβαλλοντική διάσταση. Εγώ ε, προσωπικά πιστεύω ότι είμαστε εξίσου ευαισθητοποιημένοι για τα θέματα αυτά. Βεβαίως και πρέπει να προσελκύσουμε επενδύσεις στη χώρα. Επενδύσεις όμως δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς επενδυτές και θέσεις εργασίας χωρίς εργοδότες. Ούτε και αυτό μπορεί να υπάρξει. Αλλά ούτε και ανάπτυξη χωρίς ε, να πληρούνται ε, οι απαραίτητες προϋποθέσεις όπως είναι η ανταγωνιστικότητα. Από την άλλη πλευρά βέβαια Οφείλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, όλες ε, τις επιταγές του ελληνικού συντάγματος αλλά και όλες ε, τις αποφάσεις ε, που λαμβάνονται από το Συμβούλιο Επικρατείας το οποίο είναι και πολλές φορές αρμόδιο για τέτοιου είδους θέματα. Όσον αφορά τώρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εδώ συνδέω την απάντησή μου προς τον κύριο Χρυσόγελο με την απάντηση προς την κυρία Κράτσα θέλω λοιπόν να πω το εξής. Εκτός από τα προγράμματα που αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι αρκετά αυτά και τα οποία δυστυχώς ε, δεν μπορούν να εφαρμοστούν ε, απρόσκοπτα λόγω του προβλήματος της ρεσπότητα, διότι καλούνται και οι ΜΜΕ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να συμβάλλουν κατά τη. Άρα αυτό υπάρχει, δημιουργεί πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπουν τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω του ότι, όπως σας είπα, υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Αλλά και αυτές δεν μπορούν να συμβάλλουν. Μπας περιπτώσει, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Πάντως, εκτός αυτού, εμείς ε, προσπαθούμε να ε, λάβουμε υπόψη μας τις διατάξεις ε, που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο σχετικά με το εργαλείο επιμερισμού κινδύνου και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συμφωνήσαμε σε ένα πρόγραμμα της τάξης του 1 δις με μόχλευση, όπου εκεί χρησιμοποιούμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ ως ε, εγγύηση, χέγγιο δηλαδή, για να στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα. Διαπραγματευόμεθα αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε τελικά να παρουσιάσουμε κάτι απόλυτα συγκεκριμένο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό προσβλέπουμε να γίνει το Νοέμβρη και ε, συνεχίζουμε βέβαια τις προσπάθειές μας. Τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι καλούμεθα να ε, λειτουργήσουμε μέσα σε ένα δυσίωνο, δυσμενές μάλλον, ε, οικονομικό χρηματοψηφιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί σας το είπα και στην αρχή, εδώ παίζεται η μοίρα και το μέλλον της χώρας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Αγκουράκης έχει παρακαλώ το λόγο. Of course, one minute, if I ένα λεπτό αν έχει την καλοσύνη, όχι παραπάνω. Θα είναι ελληνικό το λεπτό. Ε, κύριε Χατζηδάκη, ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Βέβαια, ε, εσείς αναφερθήκατε κυρίω στην, ε, στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνηση, η οποία πρέπει να πούμε στο Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει και την αποδοχή του ελληνικού λαού όπω ισχυριστήκατε. Αυτό εξάλλου δείχνει και οι που έχετε να περάσετε τα μέτρα στην Ελληνική Βουλή παρά το γεγονός ότι ηγείστε μιας ε, τρικομματικής κυβέρνησης. Και επίσης και τα μέτρα που έλαβε χτες η κυβέρνηση, τα απαράδεκτα μέτρα χτες στη διάρκεια της επίσκεψης της κυρίας Μέρκελ στην Αθήνα, ακριβώς αυτό μαρτύρουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά γιατί τόσο συχνά αναφερθήκατε στο πολιτικό κόστος το οποίο δεν φοβόσαστε. Ε, όσον αφορά τώρα για, το, για τον κύριο Ράιχεμπαχ, για τον οποίο τέθηκε μια ερώτηση από την κυρία Κρέλ, θα ήθελα να τη πω ότι ο κύριο Ράιχενμπαχ προχθέ εδώ στι Βρυξέλλε Προέβησε σε μια απαράδεκτη δήλωση κατά τη γνώμη μου. Είναι η επικεφαλής task force η οποία είναι επιφορτισμένη να ε, συνδράμει την ελληνική κυβέρνηση και όχι να προβαίνει σε πολιτικέ δηλώσει. Σε πάση περιπτώσει, ο κύριο η κυρία Κρέλ, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Τώρα, Ταμείο Συνοχή και ό,τι συζητήθηκε. Το βασικό ζήτημα είναι που πάνε τα χρήματα. Τα χρήματα από το Ταμείο Συνοχή πάνε βεβαίω για τι μεγάλε πολυεθνικέ. Πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε παραδείγματο χάρη στο να αυξήσει το όριο από το 6% στο 10% από τι δημόσιε συμβάσει ε, ως προκαταβολή για τι πολυεθνικές εταιρείε και φυσικά αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει εκεί που έχει οδηγήσει τη χώρα μα τώρα. Ε, δεν μπορεί κανεί να αναμένει ε, συνοχή, κύριε Χατζηδάκη γιατί ε, όλα αυτά τα χρόνια εφαρμόστηκαν πολιτικές συνοχής, έχουμε μια απόκληση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κινδυνεύει να βρεθεί η Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν πάση περιπτώσει με τις πολιτικές που εφαρμόζονται και αυτά που λέγονται περί ανταγωνιστικότητας τα προβλήματα θα ε, επιδρονωθούν ακόμα περισσότερο γιατί είναι ακριβώς το ίδιο πλαίσιο που εφαρμόστηκε όλα αυτά τα χρόνια υποτίθεται για να ε, προωθήσει τη σύγκληση και ε, φτάσαμε βέβαια στην απόκληση ε, που θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Κλείνοντα, θα ήθελα να είχατε την καλοσύνη να μα πείτε ποιοι φταίνε για αυτό το 40% μείωση που λέτε ότι κινδυνεύουν τα ταμεία συνοχής για την Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κλέμπε. Ναι, σύντομο το σχόλιο. Εδώ στο Κοινοβούλιο μιλάμε πάντα για μέτρα λιτότητας και τα συνοδεύουμε πάντοτε με τη λεγόμενο κοινωνικό σύμφωνο, δηλαδή το συνδυασμό ανάπτυξης και επενδύσεων με λιτότητα. Στη δική μας όμως Επιτροπή την Περιφερειακή είμαστε οι πρώτοι που ζητήσαμε ειδικό έγγραφο ad hoc για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που βοηθούσαν την Ελλάδα και νομίζω ότι ήταν η ταχύτερη δυνατή λύση που μπορούσαμε να βρούμε για την Ελλάδα. Αυτό το 40% που είπατε ότι θα χάσετε από τη συνοχή με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Νομίζω, ξέρω τι εννοείται γιατί και στη Σλοβενία έχουμε τους ίδιους αριθμούς αυτή τη στιγμή. Λέμε ότι θα χάσουμε 40% από την πολιτική συνοχή. Το ίδιο εννοούμε άραγε. Ευχαριστούμε. Ο Γιάννης Όλμπριχτ. Α, για τα διαρθρωτικά λέμε. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την προεσέλευσή σας συμφωνώ με αυτά που είπατε και νομίζω ότι η αξιοπιστία, η επαναφορά στην αξιοπιστία είναι το βασικότερο, είναι το πρώτο που χρειάζεται για να υπάρξει ρευστότητα και γι' αυτόν τον λόγο δεν με εκπλήσει ότι εδώ πριν από πέντε λεπτά και άλλες πολλές φορές το μήνυμα που δίνεται είναι ότι ωφελούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία οι ίδιοι που χάνουν σήμερα από αυτά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και για σας και για μας να αποδείξουμε ότι τα προβλήματα δεν οφείλονται στην πολιτική συνοχή γιατί πολλοί το λένε αυτό. Ναι. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση μεταξύ των δύο. Ερωτώ όμως, εδώ δεν ήρθατε μόνο για να εξηγήσετε ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Για μας είστε και μέλος του Συμβουλίου και γι' αυτό ερωτούμε. Θα μας στηρίξετε στο Συμβούλιο. Είστε διατεθειμένος να αγωνιστείτε για λύσεις που να συμπεριλαμβάνουν την πολιτική συνοχή, γιατί αυτό είναι το κοινό συμφέρον. Υπάρχουν δύο στοιχεία που δεν πρέπει να μπερδεύονται. Ένα, στήριξη στην Ελλάδα τώρα και μακροπρόθεσμα η Ελλάδα ως μέλος της Ένωσης που κανονικά συμμετέχει και στην πολιτική συνοχή. Για μένα αυτά συνδέονται και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μεταφέρετε στο Συμβούλιο. Εσείς ξέρετε τις λεπτομέρειες, μερικοί υπουργοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, δεν καταλαβαίνουν καθόλου την πολιτική συνοχή. Εσείς όμως ξέρετε, γι' αυτό υπολογίζουμε σε εσά, ο Γεώργιος Σταυρακάκης. Σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή που για τόσα χρόνια υπήρξατε ένα πολύ ενεργό μέλος. Ε, η ερώτησή μου ήταν και εμένα αναφορικά στην απορρόφηση των ΕΣΠΑ που απαντήσετε ήδη στην κυρία Κράτη. Σας ευχαριστώ πολύ. regards uh, the question of Mr. Πρώτα για τον κύριο Αγκουράκη. Θα ήθελα να πω ότι βεβαίως αυξήσαμε τις πληρωμές για τις κατασκευαστικές εταιρείες μέχρι 10% τις προκαταβολές. Ήταν 6% και τις αυξήσαμε στο 10% απλώς για να τις στηρίξουμε λόγω του τρομερού προβλήματος ρευστότητας. Κοιτάξτε κύριε Αγκουράκη, όταν μιλάμε για εταιρείε, μιλάμε για εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να έχουμε εργαζόμενους χωρίς εργοδότες. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε για να λύσουμε το πρόβλημα της ρευστότητας. Αν έχουμε δογματική προσέγγιση, τότε υπονομεύουμε τις προσπάθειες καταπολέμησης της ανεργίας στη χώρα μας. Κατανοώ ότι έχετε διαφορετική άποψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι και το δικό μου είναι λάθος, η εκεί μου προσέγγιση. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι με όλο το σεβασμό που σας οφείλω, η κυβέρνηση αυτή εξελέγει πριν από τρεις μήνες και εκφράζει σχεδόν το 50% της λαϊκής θέλησης. Είναι λοιπόν ισχυρή κυβέρνηση και είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να στηρίξουμε τα συμφέροντα της χώρας και των Ελλήνων πολιτών, όπως τα κατανοούμε. Όσο για το ερώτημα της κυρίας Κλίβα. Καταρχήν, ξέρουμε και εκτιμούμε την θέση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας για τις διευθετήσεις των διαρθρωτικών ταμείων για το RSI και όλα τα άλλα για την επιταχυμένη απορρόφηση για να λυθούν τα προβλήματα που θέτει η κρίση. Ανάλογα προβλήματα έχουμε και εμείς και εσείς, αλλά Εγώ αναφέρομαι στα δικά μας γιατί τη χώρα μου αντιπροσωπεύω εδώ και δεν ξεχνάω όμως αυτά που είπα και στην αρχή, δηλαδή ότι για να υπάρχει ισχυρή Ευρώπη πρέπει να έχουμε ισχυρή πολιτική συνοχής. Αλλιώς η ενιαία αγορά δεν λειτουργεί από μόνη της. Πρέπει να υπάρχει μια αντιστάθμιση με την πολιτική συνοχής. Αυτό ήταν και το όνειρο του Ιακώβου Ντελόρ και των άλλων και των ιδρυτών της Ευρώπης και αυτό πιστεύω και εγώ. Αυτό. Όλμπριχτ. Καλύψατε μερικά αυτά που ήθελα να πω. Είπατε ότι είμαι μέλος του Συμβουλίου. Δεν το είχα καταλάβει, πρέπει να σας το ομολογήσω. Γιατί αισθάνομαι μάλλον μέλος του Κοινοβουλίου. Αλλά δεν, δεν είμαι, δεν είμαι όντως είμαι τώρα μέλος του Συμβουλίου και πιστέψτε με δεν ξέχασα τι λέγαμε μαζί παλιά. Στο άτυπο Συμβούλιο της 6ης Νοεμβρίου στη Λευκοσία θα τα πω αυτά και θα υποστηρίξω φυσικά αυτές τις ιδέες και θα αγωνιστούμε όχι μόνο για τα συμφέροντα της Ελλάδας αλλά και για τη συνοχή γενικότερα γιατί αυτή είναι προϋπόθεση για να δυναμωθεί η Ευρώπη ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την κρίση. Βλέπω ότι έρχονται και άλλοι για την ψηφοφορία μάλλον. Ε. Γι' αυτό πρέπει να τελειώνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Πρόεδρο με την οποία συνεργάστηκα όταν ήμουν συντονιστής του ΕΛΚ και εκείνη ήταν επίτροπος για τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτή τη συνεργασία θα τη συνεχίσουμε και ελπίζω τελικά να έχουμε καλά και θετικά αποτελέσματα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και για την Ευρώπη στο σύνολό της που είναι ο κοινό μας οίκος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι Έχουμε εδώ και τον αρμόδιο διευθυντή από την Κομισιόν που ασχολείται με την Ελλάδα. Μπορεί να μιλήσει αλλά για ένα λεπτό το πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πράγματι λόγω του ωραρίου σας θα, δεν θα πω πολλά. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης για την παρουσίασή του και για τη σαφήνεια και ειλικρίνεια που τη χαρακτήριζε. Επιβεβαιώνω ότι ως προς την πολιτική συνοχή συμφωνούμε με αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός και οι προτεραιότητες μας είναι οι ίδιες. Η στόχη μας δηλαδή είναι η βελτίωση της εκτέλεσης ορισμένων μέτρων που έχουν συμφωνηθεί με την ελληνική κυβέρνηση και την Task Force. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να συμβάλλουμε στην ανανέωση της ροής ρευστότητας των επιχειρήσεων σε συνεργασία με την ΕΤΕ για να καταλήξουμε σε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα και τέλος τρίτη μας προτεραιότητα είναι να συμβάλλουμε όσο δυνατόν περισσότερο στην απαλοποίηση των διαδικασιών να μην αντιδρούμε πάντοτε υπό το κράτος της βιασύνης Πολλές αντιπροσωπείες πρέπει να λύσουν προβλήματα και τελειώνω λέγοντας ότι συνεργαζόμαστε στενά με τις ελληνικές αρχές για να προετοιμάσουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο και όποια και να είναι τα ποσά που θα διατεθούν τελικά σα και που ξεπερνούν τις δικές μας αρμοδιότητες θα φροντίσουμε τα μέτρα και οι χρηματοδοτήσεις που θα δοθούν να επιτρέπουν μια πραγματική αναθέρμανση της οικονομίας της Ελλάδας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ακούσετε ότι και η Κομισιόν στηρίζει αυτά που είπατε, όχι μόνο εμείς εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Συνάδελφοι, έχουμε ένα προβληματάκι. Γιατί τα καθίσματα έχουν αλλάξει για να ανταποκρίνονται στην απογευματινή συνεδρίαση με την άλλη επιτροπή. Γι' αυτό θα δυσκολευτεί η ψηφοφορία. Παρακαλώ λοιπόν τους συντονιστάς όπως τον Λαμπέρ να κινηθούν προς τη μέση εκεί της αίθουσας με την ταμπέλα των για να φαίνονται, να τους βλέπουμε κι εμείς, εμείς οι πρόεδροι, για να γίνει πιο εύκολα η ψυχοφορία. Μερικοί συντονιστές και συντονίστριες δεν αντιδρούν. Φαίνεται δεν θέλουν να μετακινηθούν. Τι να κάνουμε. Δεν Καλά. Καλά. Constanza would like to say something. Κωνσταντσα, τι θέλεις να μας πεις. Σε ευχαριστώ, Ντανούτα. Όσον αφορά στην προετοιμασία της ε, ψηφοφορίας σήμερα πρέπει να πω ότι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και θέλω να δείξω ε, τρία θέματα. Μέχρι πριν από πέντε λεπτά ε, πήραμε ε, αλλαγές για την ψηφοφορία. Αλλά δεν μπορεί κανείς να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο όταν ε, καλείται να επεξεργαστεί τόσο μεγάλο αριθμό τροπολογιών. Κατά τα άλλα, ε, δέχομαι την ε, άποψη των συναδέλφων, αλλά είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχουν οι τροπολογίες μόνο στα γαλλικά. Στο μέλλον παρακαλώ να τις υποβάλλετε και στα αγγλικά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το τρίτο που θέλω να πω και το χειρότερο για μένα είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε εδώ τρεις ή τέσσερις εκθέσεις ε, με μεγάλο αριθμό τροπολογιών που κατατέθηκαν από συναδέλφους οι οποίοι οι οποίες τροπολογίες ε, ξεπερνούν όμως την ε, δικιά μας τη δουλειά. Εχθές λοιπόν στην ομάδα εργασίας της πολιτικής μας ομάδας είπαμε ότι δεν συμμεριζόμαστε πάντα την άποψη της ε, γραμματείας. Ε, Κατονούμε βέβαια ότι είναι δύσκολο να συζητηθούν τώρα τα προβλήματα. Θα θέλαμε βέβαια να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κανόνες ή πώς ακριβώς λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Και σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορώ να φανταστώ ότι αν θέλει κανείς να έχει κονδύλια στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, ε, ίσως επιθυμεί και κάποιες διαγραφές που δεν έχουν σχέση άμεσα με την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτά ε, τα κρίνει και η γραμματεία κατά πόσον μπίπτουν οι αρμοδιότητε μα ή όχι. Σε γενικέ γραμμέ, η οχι σε γενικε γραμμε η κατασταση δύσκολη και αυτή τη φορά δεχόμεθα την απόφαση που ελήφθη ω ελήφθη γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο κατά τη διάρκεια της ε, να προβαίνουμε σε αλλαγέ. Αλλά πραγματικά θα ευχόμουν η γραμματεία στο μέλλον ε, να μπορεί να μα δείχνει έτσι και πιο παραστατικά το τι ακριβώ συμβαίνει για να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Ε, να απαντήσω, αν μου επιτρέπετε, στο τελευταίο αυτό πρόβλημα που θίξατε, που αφορά ε, στο ότι δεν έγιναν δεκτές ή στο ότι είναι απαράδεκτες ε, κάποιες τροπολογίες, γιατί... Ε, δική μου είναι η απόφαση τροπολογιες γιατι δικη μου πόσον θα δεχτώ την άποψη της γραμματείας ή όχι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια και για πρώτη φορά έχουμε ε, τόσα πολλά θέματα μαζί. Αλλά και κατά το παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις όπου ε, ψηφίστηκαν από άλλες επιτροπές θέματα δικά μας. Στην ε, συνδιάσκεψη των Προέδρων, όπου συμμετέχω και εγώ, έχουμε συζητήσει επανειλημμένα το θέμα αυτό γιατί υποβάλλονται διαμαρτυρίες από όλε τι επιτροπές. Υπάρχει ο κανονισμός 49.2 που είναι απόλυτα σαφής από αυτού και νομίζω θα πρέπει να σεβόμαστε τον κανονισμό με την έννοια ότι θα πρέπει τις ε, γνωμοδοτήσεις μας να τις στοχεύουμε μόνο σε εκείνα τα θέματα που εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε τις τροπολογίες να τις εξετάζουμε και κάτω από αυτό το πρίσμα. Αποφάσισα λοιπόν, και εδώ θέλω να με στηρίξετε, ότι ε, θα σεβαστούμε αυτόν τον κανόνα και στο μέλλον. Υπάρχει σήμερα μια κατάσταση που είναι κάπως εξαιρετική. Και πρέπει να πω ότι αρκετά καθυστερημένα αποφάσισα, τουλάχιστον αυτή τη φορά να είμαστε πιο ευέλικτοι και στο μέλλον να είμαστε έτσι πιο αυστηροί όσον αφορά στο θέμα αυτό. Υπάρχουν δύο ε, περιπτώσεις όπου μία τροπολογία είναι τόσο απαράδεκτη, είναι τόσο οφθαλμοφανές ότι κατ' ουσίαν αφορά αρμοδιότητε άλλη επιτροπής που αυτέ οι τροπολογίε δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές και αυτά τα ξεπετάει κανείς πολύ γρήγορα. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που ε, είναι αμφίσιμες και ε, ίσως σε αυτές ε, να υπάρχει κάποια έμεση σχέση με τη δική μας την Επιτροπή. Είναι ασαφές το θέμα των κόκκινων γραμμών δεν είναι σαφέ αν μια τροπολογία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ή όχι. Και εγώ αποφάσισα αυτές τι τροπολογίε να τις στείλω στι πολιτικές ομάδε, στου συντονιστέ, να αποφασίσουν αυτοί μόνοι τους. Γιατί αυτές οι περιπτώσει μπορεί νομικά να είναι σαφείς, αλλά όχι από πολιτική σκοπιά. Και να κρίνετε εσεί εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να δεχτείτε μια τροπολογία ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν έχει προκύψει η κατάσταση που έχει προκύψει σήμερα. Πάντως, στο μέλλον, εδώ συμφωνώ μαζί σας, πράγματι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι γνωμοδοτήσεις της ε, Περιφερειακής Επιτροπής να είναι καλύτερα στοχευμένες. Mm. Αυτά είχα να σας πω, κύριος Βανίστεροι. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ δίκιο έχετε πρέπει να έχουμε έγκαιρα τις πληροφορίες για να προετοιμάσουμε τις λίστες ψηφοφοριών. Αυτό το κάναμε μάλιστα χθες. Το ίδιο θα ισχύσει για την έκθεση Κρίλ και για τους άλλους συντονιστές. Την τελευταία στιγμή πήραμε τις Την Τελευταία στιγμή συντάξαμε και τις λίστες. Κάποιες φορές δηλαδή πρέπει να προσαρμοζόμαστε και μάλιστα να λαμβάνουμε υπόψη μας κάποιες λεπτομέρειες και να αλλάζουμε τις λίστες ψηφοφοριών. και κάποιες φορές θα δώσω άλλη ένδειξη ως συντηνιστής σε σχέση με αυτά που συζητήσαμε χθες, ιδίως για την έκθεση Σρέντερ για το Γεωργικό Ταμείο. Τέσσερις είναι αλλαγές α, επ' αυτού. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδίω για αυτού που είναι στο μετέχμιο. Και δεν, δεν μπορεί να προβλέψει κανεί αν θα κινηθούν προ την προς την άλλη κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, έστω και την τελευταία στιγμή, αλλά καλό θα ήταν να μα τα λέτε λίγο νωρίτερα τι είναι παραδεκτό και τι όχι, για να μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Παρακαλώ πάντω του συναδέλφου να προσέχουν πολύ καλά τι κάνει ο συντονιστή, ιδίω όταν ψηφίζουμε την έκθεση του Γεωργικό Ταμείο. Πρόεδρο, παρακαλώ ελέγξτε αν λειτουργούν οι κάρτε. Δοκιμαστικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πολλοί συνάδελφοι βλέπω ακόμη δεν έχουν ψηφίσει. Να ελέγξω παρακαλώ. Εδώ λίγη ψηφοφορία. Δύο προβλήματα έχουμε. Δύο. Κοιτάξτε, θέλω να πω, έρχεται η κάρτα μου, όπου να είναι φτάνει, γιατί χτες ε, είχαμε μια πολύ μακρά συνεδρίαση και την ξέχασα εκεί και θα μου τη φέρουνε. Άρα θα κάνετε σήμα δηλαδή, θα σηκώνετε το χέρι σας κάθε φορά. Επίσης, ένα σοσιαλιστής παραπάνω υπάρχει να μην ψηφίσει κάποιος. Τώρα είμαστε εντάξει. Θα σας λέμε όταν υπάρχουν περισσότεροι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον πιο μακρύ, πιο δύσκολο κατάλογο. Την ψηφοφορία της, εκθέσεως, της μάλλον δώσε στα άρασφαιρα γκούτα για τις άλλες υποθέσεις και την άλλη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Λοιπόν, τροπολογία 142. Υπέρ, κατά και εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι επαλήθευση της 144 άρχεται η ψηφοφορία έληξε εγκρίνεται 15 υπέρ Κατά. Τώρα επαλήθευση της 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά χές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά χές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά χές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές ε, επαλήθευση της 150. Άρχεται λίγη. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά yes Εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά ποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά ποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά ποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά ποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι επαλήθευση την τρία επαλήθευση γρήγορα όμως γρήγορα γρήγορα άρχεται η ψηφοφορία έλξη η ψηφοφορία απορρίπτεται 92 όχι 161 υπέρ 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 162 και 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 166 υπέρ. Α. Yes. Εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά 168 είπα υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά εποχές δεν ξέρω επαλήθευση Άρχεται, έλλειψη. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Όχι εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Οποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Όχι. Ξανά την 28 ηλεκτρονικά. Άρχεται λίγη. Απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά. Ξανά 177 ηλεκτρονικά. Όχι, με τα χέρια, υπέρ, υπέρ. Όχι, ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ενα υπέρ. Συμβιβαστική ενα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 260 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Ορίστε μου, ορίστε. Την 178 πριν από το, τη συμβιβαστική δεν την ψηφίσαμε. Την 178 την ξέχασα. Μάλλον την ξέχασα. Λοιπόν, 178 υπέρ πριν από, το, την, τη συμβιβαστική υπέρ κατά απορρίπτεται. Τώρα 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 184 είπαμε κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται δεύτερο τμήμα α επαλήθευση του πρώτου τμήματος ηλεκτρονικά 184 πρώτο τμήμα άρχισε η ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. 23 με κατά 20. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται Α, όχι, όχι. Δεν χρειαζόταν να ψηφίσουμε την 4. 201 υπέρ. 201 υπέρ. Γιατί 25 είχε εγκριθεί. Όχι, καταπίπτει αν δεν είχε εγκριθεί 25, αν δεν είχε εγκριθεί, αλλά εγκρίθηκε. Όχι, πώς. Όχι. Ε.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 206 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται ...207 υπέρ. Κατά. Ποιες απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά. Ποιες απορρίπτεται. 209 υπέρ κατά είχε απορρίπτεται. 210 υπέρ κατά είχε απορρίπτεται. 211 υπέρ κατά είχε απορρίπτεται. 212 υπέρ κατά είχε απορρίπτεται. 213 υπέρ κατά είχε απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά είχε εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ. Α, όχι, χωριστεί σε τμήματα η συμβιβαστική 3. Το πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής 3 υπέρ. Κατά. χές Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της συμβιβαστικής 3 υπέρ. Κατά. Παχές. Εγκρίνεται. Τώρα επιστρέφουμε στην 201 και την 32 για το άρθρο 32. 201. Ποιος είναι υπέρ της 201. Περιμένουμε, περιμένουμε. Στη σελίδα 4 είναι. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και η 32 υπέρ κατά απορρίπτεται. ...214 στη σελίδα 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 48 υπέρ, 47 λέει ομιλήτρια στη σελίδα 6. Α, είναι λάθος. Α, μάλιστα είναι λάθος. Α, είναι λάθος. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, επαλήθευση την 50. άρχισε. Κάποιος γραμμένος στη ψηφίζει εδώ πέρα, τι γίνεται. Απορρίπτεται. Λοιπόν τώρα λέει ο Φρανκ ότι κάναμε κι άλλο λάθος. Πρέπει να ψηφίσουμε για τη 48 γιατί την είχα πει 47. Την 48. Ήταν λάθος, λάθος στον κατάλογο ψηφοφορίας λοιπόν. Ξεχάσαμε τη 47. Θα διορθώσουμε, θα διορθώσουμε. 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ορίστε. Τώρα επανερχόμαστε στην 90. όχι 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 167 με προφορική τροποποίηση του συντάκτη. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροποποίησης. Όχι ψηφίζουμε λοιπόν με αυτή την προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται. 217 υπέρ. Κατά. Ποιες εγκρίνεται. Αν δεν απατώμε. Θέλετε έλεγχο. Όχι λοιπόν. Αν θέλετε έλεγχο να φωνάζετε. Έλεγχο 218 υπέρ. Τώρα είναι πολύ αργά, δεν γίνεται τώρα. 217, άντε καλά, 217 έλεγχος. Για τους Γάλλους το κάνουμε, μην το ξεχνάμε. Έληξε, εγκρίνεται. 218 συνάδελφοι, σε κάθε ψηφοφορία κάποιοι δεν ψηφίζουν ή κάποιου η μηχανή δεν δουλεύει. Πρέπει να το διορθώσουμε. Λοιπόν, 218 υπέρ. Κατά. Τα ίδια με πριν. Εγκρίνεται λοιπόν. 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 221 221 υπέρ α όχι καταπίπτει 223 ε, ε, ε. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 και 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 228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 Πάλι έχουμε περισσότερους. Τι συμβαίνει εδώ ή άλλοι λιγότερους. Τέλος πάντων. Εγκρίνεται. 234 υπέρ. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69, 70 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 236 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 και 242 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται, 74 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 243 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 244 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 245 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 246 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ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 κατά εποχές εγκρίνεται 251 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 252 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 253 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 254 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 255 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 256 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 257 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Κατά τμήματα 260 πρώτο τμήμα. Πώς, πώς, ναι αυτό ρώτησα. Μου είπαν πρώτα το πρώτο τμήμα μετά το δεύτερο τμήμα. Λοιπόν ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Υπέρ κατά αποχή δεν κρίνεται. Δεύτερο τμήμα. 261 μάλλον. Υπέρ. Το δεύτερο τμήμα τι θα γίνει. Μα μου είπατε να μην ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Έτσι μου είπατε. Πρέπει και το δεύτερο. Καλά, τότε το δεύτερο τμήμα τώρα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Ορίστε. 261 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τώρα το σκεπτικό 93 και 94 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνονται. 96 σε δύο τμήματα. Α, 95 δεν ξέχασα. 95. Πώς, πώς. Ναι, 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα σε τμήματα 96, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 98 και 99 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνονται. 100 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ, και 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 όχι 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά απορρίπτεται 111 υπέρ κατά εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά Απορρίπτεται 115 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ε, πάμε, επαλήθευση, επαλήθευση, επαλήθευση. Λοιπόν, άρχισε η ψηφοφορία για την 116. Ναι, Έληξε, απορρίπτεται πανηγυρικός. Εγκρίνεται πανηγυρικός. Ναι, γιατί μερικοί δεν σηκώνουν τα χέρια τους εγκαίρους και δεν καταλαβαίνουν αν είναι υπέρ ή κατά. Λοιπόν, τώρα οι 8 υπέρ, κατά, έχεις εγκρίνεται, 117 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά εποχές. απορρίπτεται 119 υπέρ κατά εποχές. εγκρίνεται 120 υπέρ κατά εποχές. εγκρίνεται 121 υπέρ κατά εποχές. απορρίπτεται 9 υπέρ κατά εποχές. εγκρίνεται 122 υπέρ κατά εποχές. εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 όχι 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά όχι επαλήθευση, επαλήθευση για την 132 ναι, ναι, ναι. Ένα σοσιαλιστής παραπάνω. Απορρίπτεται με 26 ψήφους κατά 21. Λοιπόν, 133 υπέρ, κατά. Κατά 21 μάλλον. Επαλήθευση και την 133. Λήθευση. Έληξε. 21-25 απορρίπτεται. 11 σε τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 135 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 136 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 13 και 137 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά έληξε εγκρίνεται με 40 ψήφους υπέρ και 6 κατά και με μία αποχή. Περνάμε στη τέσσερα ψηφοφορία τώρα. Έκθεση νομοδότης, μάλλον Ραμώνα Νικόλε Μανέσκου. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών, κατευθυντήριες γραμμές. Αρχίζουμε. Τροπολογία 26, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε την 30. 30. Αν και νομίζω ότι εγκρίθηκε. Πέρας ψηφοφορίας. Σωστά τα κατάλαβα, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Την ενέδα την ψηφίζουμε. είναι αυτό smart. 34 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 10 και 35. 10 και 35 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνονται. 11 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά αποχές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 Περνάμε τώρα σε μία ακόμη μακρά ψηφοφορία. Είμαστε έτοιμοι. έτοιμοι. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ψηφοφορία της νομοδότης της κυρίας Σρέντερ. Στο μικρόφωνο, κύριε Φανλίσταλο. Είναι 21, 17, 58, 80 και 83 έχουμε μείον εμείς, αλλά βάλτε συν για το ΕΛΚ. Μιλάω, αλλά θα τα λέω και στη διάρκεια. Δεν σας ακολουθούν, λέει η πρόεδρος, ούτως ή άλλως, γιατί τους το ζητάτε τώρα. Φυσικά, δεν τίθεται συζήτηση, αλλά ε, να μην αργήσουν. Άρα ακούμε εσάς, ωραία. Ή του ΕΛΚ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Η Κωνσταντσα τι κάνει εκεί. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 21 έχουμε προφορική τροπολογία από την ησυχή Είναι κάποιος αντίθετος. Εσείς, Σικεύσκη, μάλιστα. Άρα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία, ψηφίσουμε άνευ της προφορικής. Άνευ, σου καλά, δεν τα είπα. Μάλιστα. Ψηφίζουμε την 21 χωρίς την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 κάτω τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το δεύτερο. 23 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102 δεν είναι παραδεκτή. 24 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 103. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, τι να ελέγξουμε. Το δεύτερο τμήμα της 103, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 26 υπέρ 20 κατά, άρα εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 163. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 26. Μα δεν σας βλέπω. Λοιπόν, τι θέλετε να κάνουμε, να ελέγξουμε τον 25. Εντάξει, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, 29 κατά. Βέβαια, να προσέχουμε πρέπει. Λοιπόν, 26 ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 28 έχουμε προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος αντίθετος με αυτήν την προφορική τροπολογία. Όχι, άρα ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ, μαζί με την προφορική. Κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά. Δεν πρέπει να ελέγξουμε, τι λέτε. Νομίζω ότι απορρίπτεται, δεν είναι σαφές όμως. Ψηφίζουν ηλεκτρονικά την ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται, λέει. Καρα... Δεν βλέπω καλά σήμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, 34 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα όμως μόνο ψηφίζουμε, γιατί το δεύτερο έχει αποσυρθεί. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Εντάξει. Ελέγχο 35. Γίτσες. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 27 προς 20 πάμε στην 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ, κατά, εποχές, νομίζω απορρίπτεται. Παρακαλώ, απορρίπτεται. 100, μάλλον, συγγνώμη, 38. 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 41 υπέρ, κατά Νομίζω απορρίπτεται. 43 υπέρ. Ελέγχουμε τη 41, εντάξει. Γρήγορα παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 19 υπέρ 25 κατά. Τώρα 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Άρα, επειδή είναι τα πράγματα πολύπλοκα, προσέχτε τώρα, έτσι. 47 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Νομίζω. Θέλει κανείς να το ελέγξουμε. Θέλω εγώ τέλος πάντων. Ελέγχουμε. 48. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με την ίδια περίπου διάφορα ψήφων. 109 δεν είναι παραδεκτή. Πάμε στην 50. Υπέρ. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές και αυτό απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 56 όχι, την 111. 111 υπέρ, κατά. Ελέγχουμε την 111. Άρχεται. Σοφορεί. Εγκρίνεται. Πάμε στην 56 κατά τμήματα. Είναι πρώτο τμήμα της 56. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές το Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Ε, αυτό το ελέγχουμε. 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 22 προς 21 ψήφους. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100. Τι να κάνουμε. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε. 112. Ελέγχουμε την 112. Λάμπερ, τι να κάνω, τι να σας κάνω. Απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές. Και αυτή νομίζω ότι απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ. Κατά νομίζω απορρίπτεται. Μπορούμε να ελέγξουμε όμως την 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 προς 19. 114 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Δεν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη, άρα πρέπει να ελέγξουμε την 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 25 προς 19. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 117 χωριστά. Πρώτο τμήμα πρώτον. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 121 δεν παραδεκτή. 171 υπέρ. 171 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά. Τμηματική για την 67 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 123, τι κάνουμε εδώ. Ψηφίζουμε. 123 υπέρ, κατά αποχές Απορρίπτεται. 126 πάμε. 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 131. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Υπέρ. Ε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ. 135. 135 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, νομίζω. Ευχαρίστως να ελέγξουμε, ευχαριστω Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Mm. Εγκρίνεται, 25 22. 136 υπέρ. Κατά. Εποχές. Μάλλον το ίδιο αποτέλεσμα είναι, αλλά το ελέγξουμε και αυτό. 136. Πέρασε τι mm. Θεούλη μου. Πορύφθηκε. Με μία ψήφο ναι, ναι, ναι. διαφορά. 137 υπέρ. Κατά. Εποχές. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Αμφίροπο. Ελέγχουμε. Άρχεται Λίγη ψηφοφορία. Αυτή τη φορά είναι σαφές. Το αποτέλεσμα απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Τίποτα. Δεν καταλαβαίνω σήμερα. Δεν ξέρω. Ελέγχουμε και την 138. Πέρας ψηφοφορίας. Σοπαλία. 23-23. Απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Ελέγχουμε 174. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίφθηκε πράγματι. 175. Ο ίδιος ένας ψημός να βλέπω να υπάρχει και εδώ, αλλά υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω. Ωραία. Συμφωνείτε. Πού πάμε. 176 πάμε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Νομίζω. Ελέγχουμε την 176. Μόνο στην δεύτερη έκθεση είμαστε και έχετε κουραστεί ήδη. Ε. Τι να κάνω. Λοιπόν, 20-24. Απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται. Ελιζαμπέτ φώναξες να ελέγξω. Είναι σαφές νομίζω ότι απορρίπτεται. Λοιπόν, 146 υπέρ. κατά Ελέγχουμε, ελέγχουμε γρήγορα, γρήγορα. 146. Νομίζω απορρίπτεται εγώ, αλλά... Πέρας ψηφοφορίας. Κι όμως εγκρίνεται mm. περιέργως. Λοιπόν, 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Όχι. Τι. Mm. Ελέγχουμε. 147. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 100 ελέγχουμε. Την 149 εντάξει, φωνάστε. Ναι, ναι. Ελέγχουμε. 149. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 180. Κατά εγκρίνεται. 80. Προφορική τροπολογία Τι ηγητέ. Ποιο είναι, μάλλον υπάρχει κάποιο που είναι κατά. Κύριε Σικέσκη, είστε κατά. Άρα θα ψηφίσουμε χωρίς την τροπολογία την προφορική. Την 80. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω. Για μισό λεπτό να δούμε. Ψηφίζουμε την 153. Το έλεγξε δίπλα εδώ η Χέλα. Δεν εγκρίθηκε η 175 αγαπητοί συνάδελφοι. Λες ότι δεν εγκρίθηκε 175, άρα problem was if it was for the room not clear what has happened with one. Με την 152 πάλι είχαμε πρόβλημα και δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα ε, να κάνουμε έλεγχο στην 152, γιατί εκεί έγινε ένα λάθος και μετά να προχωρήσουμε. Έτσι θα έλεγα. Εντάξει, 152. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα λοιπόν ψηφίζουμε τα 153 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική εύσηγμα τάφ. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ορίστε. Να ελέγξουμε. Τι θέλετε να ξαναψηφίσουμε την F. Τη συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται η συμβιβαστική. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Επιτροπής μια συμβιβαστική τροπολογία απορρίπτεται. Τι μου λέτε κύριε Φανλιστελρόι, απορρίψαμε τη συμβαστική F. Άρα πάμε και τα ψηφίζουμε όλα. Α, όχι, όχι όλα, το 82. Ποιοι είναι υπέρ, μόνο δύο ήταν, 82 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Για μισό λεπτό, για μισό λεπτό να ελέγξω την κατάσταση. Για να δούμε τι γίνεται. Με 46 τι έχει γίνει. Ωραία. Ψηφίζουμε την 181. 181. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω εγώ. Οπότε πηγαίνουμε στο 83. Υπέρ. 83 υπέρ, κατά. 83 είπα. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ 80 παρακαλώ τι θέλετε να ελέγξουμε το 84 μάλιστα ελέγχουμε πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται πάμε στο 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ Κατά. Ελέγχουμε την 156. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Πάμε στην 86 υπέρ. 86 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε και αυτό. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 24 προς 20. 157 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στα παραρτήματα. Α, γιατί καταπιπνώ όλες τροπολογίες, μάλιστα. Πού πάμε, στα ρισάιτα, στις τολικές σκέψεις. Τροπολογία 1, στα τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 158, όχι, όχι, όχι. Καθίστε να το ελέγξουμε. Τι έγινε με το 164. Δεν εγκρίθηκε κατά λοιπόν η 158. Πάμε στη 2. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. 3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για την 4 έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 4 άρχεται η ψηφοφορία απορρίπτεται το δεύτερο 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Υπέρ, 91. Καταπίπτει γιατί δεν εγκρίθηκε 164. Για την 159 μιλάω, που λέει ότι καταπίπτει αν δεν έχει εγκριθεί η 164. Άρα, τον ίδιο κατάλογο δεν έχουμε. Έτσι νομίζω. Άρα, καλά λέω να ψηφίσουμε την 91, υπέρ. Αγαπητοί συνάδελφοι, 91 παρακαλώ, υπέρ ακριβώς κάτω από την ε είναι. Στην αιτιολογική σκέψη αριθμών 21. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη που έχουν σοσιαλιστές. Είναι από χθε. Τι έγινε. Κυρία Σρέντερ, πολύ απλό. Σας τα εξηγήσω εγώ. Για το Ισάτελ 21 το βασικό πρόβλημα είναι 93 και 94. Είναι λάθος. Αν έχουν τον κατάλογο που λέει 93-94. Λέει, θα έπρεπε να λέει 91-92. Δηλαδή, ποια είναι, τα σωστή, είναι η σωστή αριθμή. Recital 21 και πρέπει να λέει 91-92, όχι 93-94. Η γραμματεία έκανε το λάθο. Προσπαθήσαμε σε πολλές ε, προηγούμενες εκδοχέ τη λίστα να το διορθώσουμε. Στην τελευταία ίσως να έχει διορθωθεί. Αν η Κωνσταντσε, λέει πρόεδρος, έχει 93-94, να ξέρει ότι είναι 91-92. Λοιπόν, 91, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τη 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε απορρίπτεται 12. Πηγαίνουμε στην 101 τροπολογία που έχουμε μια προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος κατά της τροπολογίας. Τη 13 την ψηφίσαμε. Αχ, δεν την ψηφίσαμε, την ξέχασα. Δεν μου αρέσει το 13, μάλλον γι' αυτό το παρέλειψα. Είναι λίγο γουρσούζικο, αλλά τέλο πάντων. Άντε, ας ψηφίσουμε τη 13. Τουλάχιστον ψηφίστε υπέρ όλοι. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αυτό ήθελα να αποφύγω. Το 13. Λοιπόν, θέλετε να το ελέγξουμε το 13 τελικά. Απορρίπτεται. 101. Προφορική τροπολογία έχουμε. Υπάρχει κάποιο που είναι αντίθετο. Όχι. Άρα ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14. Καταπίπτει 14. 15 τώρα όμως. Ψηφίζουμε τη 15, ψήφι υπέρ. Κατά, ποχε. εγκρίνεται και τελευταία ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται με ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, 40 ψήφους, 3 κατά. Πάμε τώρα στη δεύτερη ψηφοφορία για τη Ραμόνα. Να ξεκινήσουμε. Τι είναι αυτό? Α, για τις δημόσιες συμβάσεις. Μπορούμε να πάμε γρήγορα εδώ. Τροπολογία 77, υπέρ. Κατά, ποχές. Απορρίπτεται. 78, υπέρ. Κατά, ποχές. Απορρίπτεται. 79 και 80 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται, 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 6. Όχι, τι όχι. Μη λέτε όχι, να λέτε τσεκ. Με μπερδεύετε. Ελέγχουμε την 82. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8. 8 υπέρ. Τα αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ, ελέγχουμε την 89. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Με μικρή διαφορά, αλλά απορρίπτεται. Την 90 την ψηφίσαμε, όχι. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τι ωραία να βλέπω να φεύγουν έτσι όλες αυτές τις τροπολογίες που πάμε στη συμβαστική 4. Υπέρ, κατά εγκρίνεται. 16 τώρα. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω.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 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, πάμε σε συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Πού πάμε. 128. Υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Πού πάμε, πού πάμε. falls if compromise 7 is adopted. It's not adopted. No, or amendment not adopted. Okay, so just hang on. Exactly. You have to check. Yes, you're right. I'm right. So, so we have to vote. 136. Λοιπόν, τελικά είχα δίκιο ότι πρέπει να ψηφίσουμε τα 136. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά, Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τι κάνω τώρα που πάω. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά. Νομίζω εγκρίνεται. Αν θέλετε μπορούμε να το ελέγξουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Πού πηγαίνουμε. Κατά 548. Ψηφίζουμε. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Τη 44 πρώτα ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Ελέγχουμε, ελέγχουμε, ελέγχουμε. The vote is closed. Not, not yet. People don't vote. 23 in favor. So... Εγκρίνεται λοιπόν η 147 καταπίπτει. I vote, so that's what I'm... 147 in favor. 147 υπέρ. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε για την 147. Ψηφίζουμε. Παρακαλώ ψηφίστε. Κάτι πρέπει να επαναλάβουμε γιατί κάτι δεν πήγε καλά. Ψηφίζουμε λοιπόν. Λοιπόν, ε, θα κλείσει η ψηφοφορία, αν δεν ψηφίζετε, απορρίπτεται. Τώρα τι πρέπει να κάνω. Ε, ψηφίζουμε γιατί είναι 149 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, καταπίπτει. Η 158 υπέρ, 158 παρακαλώ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται ή 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 164 και 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατάποχες απορρίπτεται. Η 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 171 υπέρ κατά, συγγνώμη, μήπως μπορούμε να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για την 171. Λαμπέρ, πώς πρέπει και εγώ να ψηφίσω. Απορρίπτεται η 171. Η 172 και 173 από κοινού, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές νομίζω απορρίπτεται. Η 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται η 174 και 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 178 και 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 και 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 και 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 184 και 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι 186 και 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, οι 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, οι 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Οι 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Οι 191 και 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 50 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 193 καταπίπτει, 54 υπέρ κατά εγκρίνεται, 55 υπέρ εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στις παραθέσεις ε, στα εκτιμώντες μάλλον 57 εκτιμώντες λέει η πρόεδρος 57 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 1 υπέρ εγκρίνεται η 61 υπέρ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 ε, η 44 δεν εγκρίθηκε κατά πίπτη. Η Κάρα λέει ότι λόγω του ότι εγκρίναμε την 44 Τώρα δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε, πρέπει να ψηφίσουμε μόνο. Ε, ποιος είναι υπέρ των τριών που δεν τροποποιήθηκαν προφορικά, παρακαλώ. Κοιτάξτε, η 44 εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Κατόπιν τούτου, εδώ δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για μια προφορική τροπολογία χωρίς την ε, προφορική τροπολογία. Υπέρ λοιπόν τώρα εγκρίθηκε, υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίθηκε. Καταπίπτει, πάμε στην 69, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα για την 71, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 4 υπέρ κατά αποχές, νομίζω ότι εγκρίθηκε, η 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε, η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα για το σύνολο της γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Έκλεισε λοιπόν η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε 32-9 είναι το αποτέλεσμα. Dear colleagues, now unfortunately have to... Συνάδελφοι, τώρα πρέπει να σταματήσουμε την ψηφορία γιατί ήδη περιμένει ο, ο προσκεκλημένος μας. Ε, θα ξαναψηφίσουμε, θα ξαναρχίσουμε στις 4.30. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε την ψηφοφορία στις 4.30 Μέσα μετά τη συνάντηση Κοτέρ και τώρα θα δώσω το λόγο στον προσκεκλημένο μας. So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 Dear colleagues, I would like to start the meeting. Συνάδελφοι, παρακαλώ, θέλουμε να αρχίσουμε. Θέλουμε να αρχίσουμε. Όσοι θέλουν να έχουν ιδιωτικές συζητήσεις, παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα ηρέμως. Καλωσορίζουμε τον Φαμπρίτσιο Μπάρκα, που θα τον γνωρίζετε από προηγούμενες συναντήσεις και που προσφέρθηκε να έρθει να μας πει πως έχουν τα πράγματα στην Ιταλία. Θα μας άρεσε να ακούσουμε ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις για τις προσαρμογές. Παρακαλώ λοιπόν τον κύριο Υπουργό Βάρκα να μας πει να κάνει την εισήγησή του. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά έρχομαι ενώπιόν σας. Νίκο. Θα σας πω μερικά πράγματα για την καλύτερη δαπάνηση, better spending δηλαδή. Μερικά αγγλικά, μερικά ιταλικά. Μια στιγμή τώρα να σβήσω το τηλέφωνο μου εδώ. Ε. Δεν σβήνει, Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο. Όχι μόνο για να αποφασίσουμε πού πηγαίνουν τα λεφτά, αλλά και πώς θα δαπανηθούν. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Better spending είναι κάτι που είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι μόνο ένα σύνθημα, γιατί όλα τα συνθήματα τελικά καταναλώνονται και δεν καταλήγουν πουθενά. Εμείς θέλουμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, δηλαδή η εφαρμογή ορισμένων κανόνων που έχουν ήδη συμφωνηθεί και πώς εφαρμόζονται αυτοί. Πρώτον, αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, υπήρξε ο συμβιβασμός του τελευταίου, της τελευταίας διάσκεψης Συμβουλίου Υπουργών. Προς έχουμε το άρθρο 87 και συζητήσαμε μια καλή λύση για να γίνει το πρόγραμμα λειτουργικό με πράξεις, με δράσεις και επίσης πολύ σημαντικό στο 87 είναι η παραπομπή που γίνεται σε αποτελέσματα σε βιωτικό επίπεδο, σε ποιότητα ζωής. Δεν βλέπετε. Α, λυπάμαι. Γι' αυτό. Τέλος πάντων. για να δούμε τα θέματα, τη συγκέντρωση των θεμάτων και των στόχων. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε δύο καλά νέα και ένα προβληματικό. Φαντάζομαι ότι μια καλή εξισορρόπηση της συγκέντρωσης και της επικουρικότητας, όπως θέλετε πέστε το, έχει επιτευχθεί από την στόχευση των προγραμμάτων 80 ή 60 τουλάχιστον της 100 και δεν θα ήθελα αυτά να αποδυναμωθούν, να νερωθούν. Είναι ένας καλός συμβιβασμός γιατί δεν λέει στην κάθε χώρα που ακριβώς να συγκεντρώσει τα κονδύλια της. Δεύτερον, επίσης είναι καλή λύση το μήνυμα που δόθηκε για το double marking. δηλαδή πρώτον όλοι οι πόροι για τους στόχους 8, 9 και 10 απασχόληση των νέων κλπ. Και το 20% μετά του Κοινωνικού Ταμείου για την κοινωνική ολοκλήρωση, συμπερίληψη. Αυτά είναι θετικά. Δεν είμαι όμως τόσο σίγουρος για το Περιφερειακό Ταμείο, το ERDF, γιατί νομίζω ότι εδώ προβλέπεται πλήρης προκαθορισμός των στόχων. Ενώ εγώ θεωρούσα ως σωστή λύση να επιλέξουν οι χώρες μόνες τους. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Τέλος. Μέχρι τώρα νομίζω ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθη είναι ο καλύτερος δυνατός για τους στόχους που προβλέπουμε, αλλά η αναλογικότητα δεν πρέπει πια να είναι δόγμα, γιατί το κατά πόσον έχουμε σωστές αποφάσεις ή τα σωστά όργανα δεν καθορίζει πόσα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν τα αυτόματα. Να μην είναι δόγμα λοιπόν η αναλογικότητα. Δεύτερος τομέας. Οι τομείς όπου θεωρώ ότι πρέπει να βελτιωθούν οι κανόνες. Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχει ακόμη τελειώσει η συζήτησή του στο Συμβούλιο, χρειάζεται ενδυνάμωση. Προς στιγμήν φαίνεται σαν κάτι κενό τελείως. Δεν είναι σαφές δηλαδή ποια είναι η στρατηγική για την συνοχή εκεί πέρα, περιφερειακή τουλάχιστον, είναι λίγο ανησυχητικό. Φαίνεται να λέει ότι η πολιτική συνοχή δεν έχει τους στόχους που θα έπρεπε. Για τις εταιρικές σχέσεις Το θέμα είναι σημαντικό του Ευρωπαϊκού Κώδικα Συμπεριφοράς για να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα θα συντάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η γνώση των συμβαλωμένων. Όσο για το την αποτελεσματικότητα του προγράμματος Performance Framework χρειάζονται ακόμη βελτιώσεις. Τέλος η προσθετικότητα. Νομίζω είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη με την απλοποίησή της και με τη σύνδεσή της με το σύμφωνο σταθερότητας. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή όλοι τα ίδια μέσα και έτσι όλοι οι πολιτικοί τα ίδια να διαθέτουν. Τέλος, δύο καινούργιοι κανόνες που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί. Υψηλού επίπεδου πολιτική συζήτηση και εξέταση. Στην νεαρινή Σύνοδο νομίζω πρέπει να εξεταστούν οι τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής της Ένωσης. Ελπίζω στο δεύτερο τμήμα να σας δείξω ότι το ίδιο το γεγονός ότι το, η συνεδρίαση για το ευρώ του Οκτωβρίου έστειλε ή θα στείλει πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα Έπειτα η ανοιχτή συνοχή. Νομίζω ότι υπάρχει ένα έγγραφο που θα ζητήσει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 16 Οκτωβρίου που θα συμπεριλαμβάνει μερικές αλλαγές του άρθρου 105 για την επικοινωνία. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση η εποπτεία και αξιολόγηση να μην αφορά μόνο ορισμένους ειδικού, αλλά όλους τους πολίτες. Και έρχομαι τώρα στην Ιταλία. Είχα έρθει και άλλη φορά να σας πω το πρόγραμμα της Ιταλίας και τώρα θα σας πω τι κατάφερε να πετύχει. Τα λέω στα Ιταλικά τώρα. Η Ιταλία έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια σε όλους τους ε, τομείς ε, στους οποίους αναπτύσσει δραστηριότητε η κυβέρνηση. Κατόπιν τούτου, φαντάζομαι δεν σας εκπλήσει το γεγονός, βλέποντας αυτό το γράφημα, ότι δεν είναι αλήθεια ότι η Ιταλία ήταν πάντα ε, η πιο σπάταλη στην Ευρώπη. Το κόκκινο, η κόκκινη καμπύλη δείχνει τα ποσοστά δαπανών ε, και η μπλε καμπύλη δείχνει την περίοδο 2000-2006 και το 7-13 είναι η κόκκινη. Το Δεκέμβριο ε, του 2011 ήμασταν στο 40% πριν από 7 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Ε, το 7-13 πρέπει να αντιμετωπιστεί για την Ιταλία ως μια ανώμαλη περίοδος ε, καθότι αυτή η περίοδος γενικότερα χαρακτηρίζεται από ανομαλίες. Αυτή η πενταετία της Ιταλικής ιστορίας. Τι συνέβη? η προηγούμενη κυβέρνηση, όχι η δικιά μας, η προηγούμενη αντέδρασε σε αυτή την κατάσταση και τον Οκτώβριο του, ε, στις 26 Οκτωβρίου ο Μπερλουσκόνη κατέθεσε ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μία πρόταση η οποία έγινε από, και από αυτή την πρόταση ξεκίνησε και από μένα προέκυψε ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο αποτελείται από συνεργασία, ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σημαίνει δηλαδή ε, περιορίζονται οι χρόνοι της δράσης, ε, μεγαλύτερη παρουσία και των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όσον αφορά τις μεμονωμένες περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει δύο task force στις δύο πιο προβληματικές περιοχές του Νότου της Ιταλίας. Σημαίνει επίσης ότι ορίζονται εθνικοί στόχοι, οι οποίοι στόχοι αυτοί αυτή προστίθενται στον στόχο νη συν η σταδιακή μείωση της συγχρηματοδότησης και στα τέλη Οκτωβρίου ε, θα φτάσουμε τα 8 δις. Τίτε λοιπόν εδώ το εξής ερώτημα. Άρα δηλαδή η Ιταλία αποδυνάμωσε ουσιαστικά την κοινοτική πολιτική. Προφανώς όχι. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, η Ιταλία ήταν η χώρα εκείνη η οποία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Η εθνική συμμετοχή στην Ιταλία ανήρχεται σε 53% του ε, συνόλου της δαπάνης ενώ 31% είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Γερμανίας 40%. Άρα δηλαδή με τη μείωση της ε, συγχρηματοδότησης η Ιταλία περνάει από το 53% στο 47%. Ακόμα δηλαδή είμαστε πολύ ψηλά ε, όσον αφορά τα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Μετά τα 8 δις αυτά παρά τις ε, ανάγκες που είχε το κράτος στην Ιταλία, αυτά τα 8 δις ε, επενδύθηκαν με δράσεις που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα πρόγραμμα δράσης, το περίφημο Action Plan. Δηλαδή δεν αφαιρέθηκε ούτε ένα ευρώ από την ανάπτυξη. Αυτά τα κονδύλια αναδιαρθρώθηκαν, ανατοποθετήθηκαν με βάση τις προτεραιότητες και κάτι άλλο. Εμείς επωφεληθήκαμε από αυτό το πρόγραμμα δράσης, από αυτά τα 8 δις, επωφεληθήκαμε για να μπορέσουμε να προκαταλάβουμε ε, την εισαγωγή κάποιων κανόνων, όπως είναι η εστίαση στο αποτέλεσμα, οι πιο ε, στενές συνεργασίες, open government και open data. Τώρα, θα αναφερθώ ε, σε κάποια αποτελέσματα. Όσον αφορά τα λειτουργικά προγράμματα, ή το λειτουργικό πρόγραμμα. Αυτό δεν είναι το πρόγραμμα δράσης, είναι τα καθημερινά προγράμματα. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει αδυναμία της Ιταλίας. Έχουμε τα στοιχεία του Δεκέμβρη του 2011. Και βλέπετε εδώ, δεν ξέρω αν βλέπετε βέβαια, τέλος αν βλέπατε θα βλέπετε ε, τον τελευταίο αστερίσκο του Δεκεμβρίου του 2012 που λέει νη συν οι δύο προηγούμενοι αστερίσκοι του Οκτωβρίου και του Μαΐου είναι οι εθνικοί στόχοι. Εθνικοί στόχοι τους οποίους ε, εισαγάγαμε εμείς για να μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο επιβάλλοντας εθνικές κυρώσεις. Βλέπετε την πράσινη γραμμή, την καμπύλη αυτή, το στοιχείο του Μαΐου ε, και εμεί νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε και τον εθνικό στόχο του Οκτωβρίου, δηλαδή το νησιν 2 του Δεκεμβρίου. Πρόκειται ε, για ένα πολύ ε, επίπονο εγχείρημα. Αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το πρόγραμμα δράση. Αυτά τα περίφημα 8 δις. εδώ είναι ένα λάθος. Λέει 9,4. Δεν είναι 9,4. Είναι 8 τα δις. Και βλέπετε εδώ τις προτεραιότητες. Ε, Προτερότα είναι οι νέοι, όπως ε, πολύ σωστά ε, μας είχε πει και η Επιτροπή και το Συμβούλιο, μέσα από την παιδεία, την κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, την μέρημνα για τα παιδιά και τη δικαιοσύνη. Προβλέπονται και άλλες δράσεις για τους νέους, αλλά προβλέπονται και κάποιες νέες παρεμβάσεις κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και προβλέπεται και περιορισμό του χρόνου εκδίκασης δικαστικών υποθέσεων. Υπάρχουν και παρεμβάσεις ε, στις επικοινωνίε και στις ε, μεταφορές, σιδηρόδρομοι, ψηφιακό θεματολόγιο και υπάρχει και ένα στοιχείο που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα. Εδώ προβλέπεται και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, οι περίφημες ευφυείς πόλεις. Εδώ ε, από το 2014 έως το 2020 προβλέπεται μια συγκεκριμένα στρατηγική για αυτές τις ευφύς ε, πόλεις. Εμείς όμως προτρέχουμε, ε, αυτό αφορά κυρίως τον, την Υπουργό Παιδείας. Επίσης θέλω να πω ότι η αναχρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκε και για να σωθούν κάποια προγράμματα τα οποία δεν προλάβαιναν να ολοκληρωθούν στις 31 Δεκάτου του 2012. Νομίζω ότι έχω τελειώσει. Φτάνω τώρα σε κάποια επιτεύγματα. Ε, το πρόγραμμα της παιδείας ε, που είναι το μεγαλύτερο πρόκειται για 1,4 δις. Το πρόγραμμα αυτό από τον Δεκέμβρη, τον προηγούμενο Δεκέμβρη, έχει ήδη απαιτήσει το 70% των ιδίων πόρων. Ε, εκεί θα επενδυθεί ήδη το 70% των ιδίων πόρων. Επίσης, εισήχθη ένας ειδικός φόρος για τους μειονεκτούντες εργαζόμενους. Ε, η απήχηση σε αυτό το διαγωνισμό ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Είχαμε ε, μία απάντηση για πάνω από 300.000 300 ε, εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, για τη δικαιοσύνη, ξεκινάμε μετά από πέντε μέρες το πρόγραμμα και θα αφορά την ICT, την πληροφορική την εισαγωγή της στην Ιταλία. Γιατί ας πούμε στο νότο της Ιταλίας για τις επιχειρήσεις ο χρόνος που χρειάζονται για την εκδίκαση υποθέσεων είναι τετραπλάσιο, πενταπλάσιο από ό,τι στη Βόρεια Ιταλία. Όσον αφορά τους νέους, υπάρχουν πολλά και μεμονωμένα προγράμματα. Αν θέλετε, πολύ ευχαρίστως ε, να απαντήσω στο έτοιμά σας ε, τι είναι αυτό το Messenger. Είναι ένα τελευταίο πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Μετά για το ψηφιακό θεματολόγιο μπορείτε να δείτε στην διαφάνεια. Έχουν ήδη εγκριθεί ε, κάποια σεμινάρια στις Βρυξέλλες για τους σιδηρόδρομους. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Η Ιταλία είναι μια χώρα που έχει πρόβλημα να δρομολογήσει μεγάλα προγράμματα γιατί υπάρχει κάποια ε, σχέση ανάμεσα σε ε, θεσμούς ε, και πολίτες. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια νέα μορφή συνεργασίας στη διαδρομή Νάπολη-Μπάρι. Εκεί βρίσκεται το 55% της βιομηχανίας της Ιταλίας το να ε, περιορίσει κανείς τις 3,5 ώρες σε 48 περίπου λεπτά, αυτό καταλαβαίνετε είναι κάτι το πολύ εντυπωσιακό. Μετά υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα ε, που ήδη το είχε πει ο κύριος Χάνκ στην προηγούμενη κυβέρνηση και ελπίζουμε για αυτό το πρόγραμμα ο Επίτροπος να μπορέσει να διεπιτόπου τα πρώτα στάδια εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Και περνάω πάλι στα αγγλικά. Το σχέδιο ανάκαμψης της Ιταλίας θα το περιγράψουμε και σήμερα σε μια διάσκεψη τύπου, θα το παρουσιάζω και εγώ, και σε, ένα, σε μια ιστοσελίδα που μπορείτε να τη συμβουλευτείτε και συμπεριλαμβάνει όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 414 δισεκατομμυρίων ευρώ και συμπεριλαμβάνει επίσης προγράμματα που χρηματοδοτούνται και από την Ιταλική Περιφερειακή Πολιτική, παραδείγματο χάρη. αυτό το πρόγραμμα για την Νεάπολη για το μετρό είναι επιτυχές, υπάρχουν όμως εκατοντάδες που δεν είναι και τόσο επιτυχή και τα δείχνει όλα η σελίδα Τι δαπανάτε, πώς δαπανάτε και κάθε τρεις μήνες ενημερώνεται η σελίδα, μπορεί να τη δουν όλοι οι πολίτες. Οι φοιτητέ, οι αναλυτές, τα πανεπιστήμια, να δουν αν οι δεξιοί δήμαρχοι τα καταφέρνουν καλύτερα από τους αριστερούς ή όχι, Ό,τι θέλουν μπορούν να δουν, ό,τι θέλουν. Έτσι έχουν μάτια οι πολίτες στην διοίκηση. Και 14.000 ήδη το έχουν δει και απ' έξω από την Ιταλία. Και ήδη έχω δει αποτελέσματα διοικητικά. Όλοι καταλαβαίνουν ξαφνικά ότι η δουλειά των ανωνύμων δημοσίων υπαλλήλων παρακολουθείται αυτή τη στιγμή από όλους και γι' αυτό βελτιώνεται η δουλειά τους ξαφνικά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βάρκα. Όποιος θέλει να μιλήσει παρακαλώ να μου το λέει, να σηκώνει το χέρι του. ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, κάποια ε, παρατηρήσεις για δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα ε, το σύστημα και μετά για την Ιταλία. Σε ό,τι αφορά το σύστημα, αυτό το οποίο γενικότερα στο σύστημα αλλά και στη δική σας ομιλία προξενεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η θεματική συγκέντρωση. Το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη για συγκέντρωση. Το ερώτημά μου όμως είναι πώς δημιουργείται αυτή η θεματική συγκέντρωση και πώς μπορούμε να καταστήσουμε πιο ευέλικτο το σύστημα από πλευράς ε, επικορικότητας. Αλλά από πλευράς συγκέντρωσης δεν έχουμε καταφέρει να είναι το ίδιο ευέλικτο. Πρέπει και το Συμβούλιο να καταλάβει ότι εμείς αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι ε, τα κράτη-μέλη να τα υποχρεώσουμε κατά κάποιο τρόπο σε μεγαλύτερη ε, συγκέντρωση. Αλλά χρειάζονται περισσότερα περιθώρια. Κάτι που δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο αλλά μάλλον έγινε πιο ξεκαθαρό μετά τη δική σας όμιλη, είναι πού επικεντρωνόμαστε τελικά ε, στο κοινωνικό ταμείο και πού επικεντρώνουμε το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρέπει να δούμε τα μηνύματα, νομίζω στα 11 αυτά. Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό ε, ταμείο, σε ό,τι αφορά το μάλλον το CSF, τι προτείνει η Κομισιόν. Προτείνει να υπάρχουν κάποιες δράσεις, αλλά υπάρχουν και οι προτεραιότητες επενδυτικές. Άρα δεν μπορούμε να αναφέρουμε δύο φορές τι πράγματα στο έγγραφο. Με ποια συνέπεια. Αν έχουμε στις επενδυτικές προτεραιότητες, τότε στο CSF θα είναι διαφορετικές οι προτεραιότητες. Τι, στρατηγική ή συγχώνευση των ταμείων που είναι η στρατηγική εξόδου. Το CSF δηλαδή, το κοινό, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, ε, αυτή την, ε, το σκοπό να έχει. Βέβαια, από την αρχή η Κομισιόν λέει κατεξουσιοδότηση εν πράξεις. Ε, το ξεκαθαρίσαμε, δεν θα είναι κανονισμοί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τι είδους δράσεις, γιατί είδους δράσεις μιλάμε. Και το ερώτημά μου σε ό,τι αφορά την Ιταλία. Ίσως να μην τα λέω καλά τα νούμερα, να μην καταλαβαίνω καλά τι θα πει συγχρηματοδότηση, αλλά τι κρύβεται πίσω από τα διάφορα, διαφορετικά επίπεδα εθνικής συγχρηματοδότησης, γιατί έχουμε κανόνες. Έτσι δεν θα έπρεπε να τηρούνται οι κανόνες. Ε, τέλος πάντων, μπορεί να φταίει το γεγονός ότι είμαι αδαής για το θέμα αυτό. Ε, κύριε Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήθελα να κάνω τις εξής ε, δύο-τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, κύριε Υπουργέ, και η χώρα σας όπως και η Ελλάδα αλλά και γενικότερα η Ευρωζώνη βρίσκεται σε μια παρατεταμένη, ε, βρίσκεται σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση Ιταλία, Ελλάδα, Νότος, αλλά γενικότερα η Ευρωζώνη και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία αυτή η οικονομική κρίση θα συνεχιστεί τουλάχιστον τα, ε, τα επόμενα δύο με τρία χρόνια. Ε, χειριζόσαστε ένα πρόγραμμα για το Ταμείο Συνοχής ε, το οποίο δεν ξέρω σε τι βαθμό παίρνει υπόψη της αυτό το στοιχείο της κρίσης. Από τα στοιχεία που παρουσιάσατε η εντύπωσή μου είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που χρησιμοποιείται από το Ταμείο αυτό προορίζεται κυρίως να αμβλύνει τις αντιδράσεις του κόσμου, των νέων, των εργαζομένων, αυτών που υποφέρουν περισσότερο από την κρίση, από ότι να βγάλουν τη χώρα σας ε, από το πρόβλημα. Και χωρίς μια ανάπτυξη, και κυρίως μια ανάπτυξη της βιομηχανίας κατά τη γνώμη μου και άλλων τομέων, Ούτε στην Ιταλία και ούτε στην Ελλάδα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Με αυτή την έννοια, ενδεχομένως εγώ δεν κατάλαβα καλά. Κάνατε λόγο για το γεγονός ότι όσον αφορά το κοινό στρατηγικό πλαίσιο υπάρχουν κάποιες ασάφειες ή ακόμα δεν είναι ξεκαθαρισμένα πλήρως ποιο είναι αυτό το πλαίσιο. Αν εγώ καταλαβαίνω καλά και διαβάζω τα κείμενα, σχεδόν αποκλειστικά το, κοινο, το, το πλαίσιο καθορίζεται από την Ευρώπη 2020. Λοιπόν, ε, αυτό το κοινό στρατηγικό πλαίσιο είναι σίγουρο ότι για χώρες σαν τις δικές μας θα, θα οξύνει ακόμα περισσότερο την απόκληση που έχουν από τις αναπτυγμένες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ απλά γιατί δεν έχουν τις προϋποθέσεις, τουλάχιστον την Ελλάδα είναι σίγουρο αυτό, να, ε, να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, Κλείνοντας, ε, ήθελα την άποψή σας σε σχέση με αυτό, το ζήτημα πώς δηλαδή η Ευρώπη 2020 μπορεί να ενταχθεί στα επιλογές σας και ένα δεύτερο, αν υπάρχει μια εκτίμηση στην Ιταλία για το πού επιστρέφουν ε, τα κοινοτικά ποσά. Θα, για να σας βοηθήσω σας πω το εξής. Ο κύριος Χάν, ο Επίτροπος Χάν, είχε μιλήσει ότι στην Πορτογαλία για κάθε ένα μάρκο που πάει στην Πορτογαλία τα 85 επιστρέφουν στη Γερμανία. Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι το 40 με το 45% των ε, επενδύσεων από τα ταμεία συνοχής επιστρέφουν στις χώρες τους δότες. Στην περίπτωση της Ιταλίας ποια είναι η αναλογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, please. Ευχαριστούμε κυρία Ματσόνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες ε, ερωτήσεις ε, σχετικά με αυτό το θέμα των δύο μερών που είπατε στην παρέμβαση σας. Όσον αφορά λοιπόν στην βελτίωση των δαπανών, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν είναι σαφή για μένα. Κυρίως όσον αφορά στην ε, αιρεσιμότητα εξάντε. Δηλαδή, μιλάμε για προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται εκ των προτέρων για να ε, προσανατολιστούν οι επενδύσεις. Μιλάμε για όρους και προϋποθέσεις που αφορούν σε όλες τις χώρες. Είναι στάνταρτ αυτές οι προϋποθέσεις. Και ε, όσον αφορά αυτό το θέμα, εγώ παρουσίασα τροπολογίες που έχουν ως στόχο να έχουμε κατά νου μια μορφή ευελιξίες η οποία θα μπορούσε να λάβει υπόψη στο το σημείο εκκίνησης ε, της κάθε χώρας. Γιατί η πολιτική συνοχής ε, φιλοδοξεί στο να καλύψει το κενό που υπάρχει. Όμως αυτή η θεωρία της πολιτικής συνοχής ε, πολλές φορές στην πράξη φαλκιδεύεται διότι όταν καθορίζονται οι κανόνες τελικά δεν λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει διαφορετικό σημείο εκκίνησης. Εγώ αυτό, μάλλον δεν κατάλαβα από την ε, παρέμβασή σας. Είσαστε υπέρ αυτού ότι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι στην πολιτική συνοχή τελικά δεν ξεκινούν όλοι από την ίδια αφετηρία και να ληφθεί αυτό υπόψη και στον επόμενο προγραμματισμό όσον αφορά τώρα την απόδοση. Και εδώ ανησυχούμε γιατί πολλοί Ιταλοί συναντέλφοι ε, παρουσίασαν μια τροπολογία ε, όπου γίνεται λόγος ε, για όλο και μεγαλύτερη γραφειοκρατία σε αυτήν την Επιτροπή. Γιατί εμείς είχαμε καταθέσει μια συμβαστική ε, τροπολογία η οποία ε, δεν αφορούσε το εκπαιδευτικό στοιχείο της παρέμβαση. Εμείς πιστεύουμε ότι όποιο κάνει λάθο θα πρέπει και να πληρώσει. Δηλαδή οι χώρε που δεν σέβονται του κανονισμού ε, θα πρέπει πράγματι να πληρώνουν. Αλλά σε αυτό το τομέα οι κυρώσει ε, θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή να έχουν ως στόχο τη βελτίωση. Κατόπιν τούτου εμεί ε, καταθέσαμε αυτή την τροπολογία η οποία επανεμφανίστηκε με συμβασμό για να καταργηθεί το τέταρτο κόμμα του 20 κατά τη διάρκεια της ε, ψηφοφορίες Τελικά η ψηφοφορία, ε, κατά τη διάρκεια της τελικά ψηφίστηκε κάτι, δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς ψηφίστηκε. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει αυτό το πλαίσιο της απόδοσης, να υπάρχει στους κανονισμούς. Ε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς ότι θα πρέπει να ξεπερνιούνται τα προσκόμματα της γραφειοκρατίας. Όσον αφορά τώρα τη σωρευτικότητα, την προσθετικότητα, εσείς είπατε ότι δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή καμία εξαίρεση. Δεν το κατάλαβα όμως αυτό. Τι μήνυμα θέλετε να περάσετε. Λαμβάνοντας υπόψη και αυτά τα οποία έχουν λεχθεί και αυτά που προκάλεσαν οι παρεμβάσεις του συναδέλφου Όλμπριχτ. Θα λοιπόν λιγάκι να μας ξεκαθαρίσετε. Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η προσθετικότητα σε σχέση με την Ιταλία και τις άλλες χώρες. Όσον αφορά τώρα την Ιταλία, στο δεύτερο τμήμα της ε, παρέμβασής σας και εγώ κάποια θέματα δεν τα κατάλαβα. Εσείς αναφερόμενος πολύ σωστά ε, σε αυτά που έλεγαν χώρα όταν η προηγούμενη κυβέρνηση ζήτησε να υπάρξει μια ενισχυμένη συνεργασία δηλαδή τον ορισμό ενός προγράμματος ε, το οποίο ε, θα προέβλεπε συντονισμένες ενέργειες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αναφερόμενος στα στοιχεία προσθέσατε την ικανοποίησή σας και είπατε ότι είσαστε ικανοποιημένοι γιατί έχουν επιτευχθεί στόχοι που καταρχήν είχαν οριστεί για το Μάιο. Εγώ δεν θέλω να έρθω σε σύγκρουση μαζί σας, θα πω όμως αυτά που διάβασα στον τύπο. Ο εθνικός μας τύπος ε, μιλάει για έναν υπουργό ο οποίος αναφέρεται σε στόχους που δεν έχουν επιτευχθεί όχι μόνο στη Νότια Ιταλία και όχι μόνο όσον αφορά τα λειτουργικά αλλά και τα εθνικά προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να γνωρίζω ποια ακριβώς είναι η διαφορά. Είναι δύο δηλώσεις που μας ε, ανησυχούν ε, ενώ εσείς ανακοινώνετε ότι είσαστε σίγουροι ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου. Θα ήθελα να γνωρίζω τελικά τι θα γίνει στις ε, περιοχές του Νότου, κυρίως στην Καπανία, γιατί εκεί ξέρετε ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση. Εσείς λέτε ότι θα έπρεπε να υποστηριχθεί η ε, περιοχή αυτή για να επιτύχει η τοπική αυτοδιοίκηση του στόχου, ενώ ο τοπικός εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης λέει ότι ε, φταίει και τη κυβέρνηση. Μήπως μπορείτε να τελειώνετε σιγά σιγά. Κι άλλη μια ερώτηση. Εσείς ε, παραθέσατε ένα εθνικό πρόγραμμα το οποίο ε, αναδιατάσσει τους ε, πόρους, το ψηφιακό θεματολόγιο, την εκπαίδευση για τους νέους και πολλά άλλα. Και θέλω να σας ρωτήσω, Ποιες ακριβώς παρεμβάσεις προβλέπονται για, την, ε, για το ψηφιακό θεματολόγιο και για τους νέους. Και αυτό το πρόγραμμα δράσης που είναι τόσο γενικό, περιλαμβάνει τα πάντα. Και τελικά ε, δεν νομίζω ότι προβλέπετε αντίφαση με τους στόχους. Κοιτάξτε, έχουμε άλλους τέσσερις ε, που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Ένα λεπτό παρακαλώ ο καθένας, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ε, ακούσουμε τις απαντήσεις του Υπουργού. Τώρα λοιπόν, οι συνάδελφοι που θα λάβουν το λόγο, πραγματικά να μην μακρηγορήσουν, μόνο ένα λεπτό. Γιατί αλλιώς θα χρειαζόμαστε ένα κανονικό σεμινάριο για την Ιταλία, αλλά δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό σήμερα. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η παρέμβαση της ε, συναδέλφου Ματσόνη σχετικά ε, με τις αντιφάσεις ε, που υπάρχουν στο site του Υπουργείου και αυτά που μας είπατε εδώ, Αυτά δεν θα τα επαναλάβω. Αλλά ίσως μπορείτε να τοποθετηθείτε από αυτού. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε τρία θέματα. Πρώτον, συγχαρητήρια, δεύτερον, κριτική και τρίτον, ε, εξηγήσεις. Συγχαρητήρια, καταρχήν, για τις ε, γνώσεις σας και τις ικανότητές σας ε, που σας ξεχωρίζουν από τους προκατόχους και από άλλους συναδέλφους. Αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Αυτό όμως που δεν μας χαροποιεί τόσο πολύ ε, εδώ περνάω στα δυσάρεστα σε αυτή την τακτική ε, του καρότου και του μαστίγιου. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάποιες ε, ανησυχίες. Το Κοινοβούλιο για πρώτη φορά έχει τη δυνατότητα της συναπόφασης. Και σε αυτά που μας είπατε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν βαδίζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρίως όσον αφορά την ε, υποδιέρεση των περιφερειών σε τρεις κατηγορίες. Ξέρω ότι είστε υπέρ της διαγραφής ε, της μεσαίας ε, κατηγορίας γιατί έτσι θα τιμωρηθούν κατηγορίες όπως το Αμπρούτσο, η Σαρδινία. Εγώ από την προφορά μου θα καταλάβετε ότι έρχομαι από την περιοχή αυτή, από το Αμπρούτσο. Έχω την προφορά της περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν διαρωτώ με, γιατί έχετε αυτή τη στάση που δεν λαμβάνει υπόψη της την ε, θέλησή της ε, να υπάρχει αναδιάταξη των κατηγοριών. Μήπως μπορείτε να μας πείτε και λίγα λόγια για την παρέμβαση που προβλέπετε, για την πομπία. Ε, αναφέρομαι ε, στην πομπία και στο σεισμό. Αυτά είναι δύο θέματα που αφορούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να δώσετε κάποιες διευκρινήσεις. Ε, Κύριος Καρόνα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρξει κάποια διευκρίνηση για τον τρόπο με τον οποίο η νέα κυβέρνηση προτίθεται να επιληφθεί του θέματος των κονδυλίων και της πολιτικής συνοχής. Πρόκειται για ένα επίπονο εγχείρημα, έτσι χαρακτηρίζεται όλη αυτή η προσπάθεια, αυτό όμως ε, διότι τα τελευταία χρόνια δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Συμφωνώ λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν περισσότερες διευκρινήσεις από ό,τι μέχρι τώρα και να δούμε τι κατόρθωσε να επιτύχει τα τελευταία χρόνια η Ιταλία. Τα τελευταία πέντε χρόνια, είπαμε, χαρακτηρίζονται από ονομαλίες. Εγώ πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι πώς θα μπορέσουμε στα επόμενα 7 χρόνια να αποφύγουμε αυτά που έγιναν κατά το παρελθόν. Τι είδου πρωτοβουλίε προτίθεται να αναλάβει η Ιταλική κυβέρνηση. Παραδείγματο χάρη, σημαντικό είναι το πρόβλημα της ε, επικοινωνίας, της ανακοίνωσης, της ενημέρωσης περισσότερο στην, της τοπικής αυτοδιοίκησης για το τι ακριβώς παίζεται για τα επόμενα 7 χρόνια να μάθει η τοπική αυτοδιοίκηση τι θα γίνει με τα θέματα που διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να ξέρουν και αυτές να μπορούν να συζητήσουν για αυτά που θα ε, λάβουν χώρα τα επόμενα 7 χρόνια. Και επίσης, ποια είναι η θέση της κυβέρνησης όσον αφορά τη μακροοικονομική κατάσταση της χώρας. Και θα ήθελα να γνωρίζω στο τέλος του 2013 ποιο θα είναι το εθνικό ε, ποσοστό ε, απορρόφησης ε, κονδυλίων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σύντομα με ένα λεπτό που έχω στη θέση μου θέλω να ευχαριστήσω τον Ιταλό Υπουργό Δευκής Συνοχής και να του πω συγχαρητήρια για την πολύ καλή παρουσίασή του. Εγώ νιώθω ε, και εγώ φιλοευρωπαίστρα, κατάγομαι από τον Νότο και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Και αυτές οι πληροφορίες και για τη χώρα μου είναι πολύ σημαντικό να φτάσουν και στην κοινή γνώμη στους πολίτες. Θέλουμε να πάψουν να είναι αποστασιοποιημένοι και απογοητευμένοι από την Ένωση. Οι πολίτε μα και η πολιτική συνοχή είναι ακριβώ η πολιτική που του είναι πιο προσφυλή και την εκτιμούν περισσότερο. Πράγματι, πολύ σοβαρό είναι αυτό που είπατε, ότι τα προσεχή ταμεία, τα επόμενη περίοδο προγραμματισμού πρέπει να έχουν ε, έναν ισχυρό προγραμματισμό ή προϋπολογισμό, ιδίως για τις μεσαίες περιφέρειες, κατηγορίες, που αλλιώς θα υποβαθμιστούν. Πάρα πολύ σημαντική είναι η προσοχή που πρέπει να δοθεί στην Ιταλία και στις άλλες περιοχές του Νότου. Ντεάντζιλης, τελευταίος, τελευταίο λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, θα υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Ε, αναφερθήκατε εξάντε ερεσιμότητα, που νομίζω συμφωνώ μαζί σας. Θα ήθελα για λίγο να γνωρίζω και τη θέση της κυβέρνησης, δηλαδή να προσέξει η κυβέρνηση έτσι ώστε αυτή η αιρεσιμότητα να μην ε, γίνει ιδιαίτερα τιμωρητική. Θα πρέπει να υπάρχει και κάποια, κάποιες μορφής ευελιξία. Δεύτερον, όσον αφορά την πολιτική συνεχής, όπως συζητείτε αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το οικοδόμημα ε, τελικά μάλλον θα αφαιρέσει κονδύλια από τις περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές. Εγώ την αισθάνομαι αυτή την ανησυχία, γιατί σε μια περίοδο κρίσης οι περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές μπορούν να αποτελέσουν το μοχλό για να επανέλθει η ανάπτυξη, να επανέλθουν οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας. Επ' αυτού λοιπόν ε, θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός. Τρίτο ερώτημα αφορά στον πολιτισμό. Εμείς εδώ θεωρούμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι μια πολύ μεγάλη κληρονομιά και αποτελεί παράλληλα και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Παραδείγματο χάρη, στη δική μας τη χώρα η ανάπτυξη, η πρόοδος, η εργασία έχουν άμεση σχέση με τον πολιτισμό. Αλλά τι πιστεύει άραγε η Ιταλική κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γιατί τελικά δεν χρησιμοποιούνται κονδύλια για την προαγωγή αυτού του τόσο σημαντικού τομέα. Τέλος, εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δουλειά που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες. Επίπονο το εγχείρημα, όπως ε, πολύ σωστά αναφέρθηκε, αλλά θα αναφερθώ λιγάκι στην ποιότητα των δαπανών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα, δηλαδή πώς ε, τα κονδύλια επενδύονται σωστά σε παραγωγικές επενδύσεις, σε επενδύσεις που μπορούν να επιφέρουν την ανάπτυξη και κυρίως εργασία στους νέους. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Θα ακολουθήσω το ίδιο σχήμα, την ίδια σειρά των ερωτήσεων. Οι προτεραιότητες είναι το κυριότερο θέμα. Και χαίρομαι για αυτά που είπατε για την σε και συγκέντρωση. Τα είπατε πιο πιστικά και από μένα τον ίδιο. Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες για να φανεί ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερος συνδυασμός. Δηλαδή και περισσότερη συγκέντρωση και περισσότερο περιθώριο επιλογής. Χωρίς όμως να επιβάλλουμε στις περιφέρειες προγράμματα που να μην ανταποκρίνονται στη φύση τους. Ως προς το τι εννοώ όταν λέω ότι χρειάζεται το κοινό στρατηγικό πλαίσιο να μην είναι κενό περιεχομένου. Πάρτε το παράδειγμα που πήρα για την Ιταλία. Το σχέδιο δράσης της Ιταλίας είναι μήπως υπερβολικά ευρύ. Όχι. Γιατί η συγκέντρωση δεν αφορά, δεν σημαίνει να κάνουμε πολλά πράγματα του ίδιου τύπου, αλλά να υπάρχει μια στρατηγική που έχει κάποια περιφερειακή βάση. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε 5, 6, 7 διαφορετικούς τύπους, αλλά έχουμε στρατηγική ή όχι. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε, δεν έχω όμως το χρόνο να σας την περιγράψω. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, να τα ξαναπούμε άλλη φορά. Για μας θα ήταν πολύ καλό, γιατί χρησιμοποιούμε το σχέδιο δράσης ως υπόδειγμα για την περίοδο 14-20 για να σας πείσουμε ότι έχουμε στρατηγική. Ένα παράδειγμα, τι θα πει κοινωνική προστασία, δεν σημαίνει τίποτα καθε αυτό, αλλά τι εννοούμε. Αναλύοντας την κατάσταση στο νότο της Ιταλίας, δεν έχει νόημα να βάζουμε χρήματα σε επιχειρήσεις, πρόσωπα, εργαζόμενους, αν δεν δημιουργούμε ταυτόχρονα μία, το αίσθημα στους πολίτες ότι εξυπηρετούνται. Γιατί στο νότο της Ιταλίας δεν παίρνει ο κόσμος αυτά που θεωρούνται φυσικά αλλού. Να υπάρξει ένα αίσθημα ηθαγένειας στο νότο. Α, ούτε αυτό όμως είναι η πλήρης απάντηση Το θέμα είναι πώς επιτυχάνεται ο στόχος. Άμα απλώς χτίσουμε σχολεία ή παιδικούς σταθμούς δεν κλείνουμε τίποτα αν δεν έχουμε μια περιφερειακή στρατηγική για όλα αυτά. Οι ίδιοι τύποι επενδύσεων μπορούν, ή μπορούν, να, μπορούν να έχουν να καλύπτονται από μια στρατηγική ή όχι και η Ένωση μας βοηθάει όχι να μπούμε σε κουτιά αλλά να δείξουμε τι σημαίνει η ύπαρξη στρατηγικής. Um, uh, Άλλα ερωτήματα. Οι προϋποθέσεις. Σε μερικές περιπτώσεις Νομίζω ότι πρέπει να παίρνουν υπόψη τους το σημείο εκκίνησης, τον τόπο εκκίνησης, σε άλλες όμως όχι. Το έχουμε δει αυτό στο νότο της Ιταλίας. Αν δεν υπάρχουν μερικές βασικές προϋποθέσεις, ας πούμε για την διαχείριση των αποβλήτων, να μην δαπανάμε ούτε δεκάρα, ενώ σε άλλες περιφέρειες πρέπει. Άρα δεν ισχύουν τα ίδια για όλες τις περιφέρειες. Η απάντηση λοιπόν είναι εξαρτάται. Συμφωνούμε απόλυτα για το γενικό στρατηγικό πλαίσιο και για την προσθετικότητα εγώ είπα ότι υπάρχει ο κίνδυνος σύμφωνα και με το Συμβούλιο να εξαιρεθούν οι μεταβατικές περιφέρειες. Αυτό εννοούσα. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να δοθούν τέτοιες εξαιρέσεις. Και τέλος, για τα συστημικά προβλήματα, τι θεωρεί η Ιταλία. Ποια είναι λοιπόν η θέση Ιταλίας ε, για τις ε, περιοχές που βρίσκονται σε μετάβαση. Πάρα πολύ απλή ότι αυτές ε, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής όπως σε όλες τις χώρες. Η Ιταλία θεωρεί ότι μπορεί να ικανοποιήσει υλοποιήσει τις ανάγκες τους μέσα από τους δικούς της ε, τους πόρους, ε, πόρους και εθνικούς ε, βέβαια και κοινοτικούς, αυτό αναμφίβολα. Άρα δηλαδή ταιριάζει στην Ιταλία το να μπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα με εθνικούς πόρους. Εγώ βεβαίως ως Ιταλός, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, καταλαβαίνετε ότι θα είμαι δυσαρεστημένος. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έχουν σχέση με την Ιταλία, υπάρχουν πράγματι διαφορές στη συγχρηματοδότηση και αυτές οφείλονται στο ότι οι κανόνες κοινοτικής συγχρηματοδότησης καθορίζουν το ελάχιστο. Και η Ιταλία έχει πάει πολύ πιο πάνω από αυτό το κατώτατο όριο. Απλά είναι τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν συνειδητοποίησαμε που πρέπει να επανέλθουμε. Γιατί Είχαμε δώσει πάρα πολλά στα κοινοτικά κονδύλια, όμως το να επανέλθουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι τα κονδύλια τα πήραμε και χαθήκανε, απλά τα τοποθετήσαμε αλλού στο πρόγραμμα δράσης. Όσον αφορά αυτή την πολύ λεπτή θέση της κρίσης, άλλα τρία λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Θα τα αφήσω αυτά τη κρίση για το τέλος. Για την κρίση λοιπόν θέλω να πω το εξή. Πράγματι έχετε δίκιο, η Ιταλία έχει λάβει υπόψη στην κρίση και αυτό φαίνεται κυρίως σε επιλογές τις οποίες κάνει. Παραδείγματος χάρη έχει λάβει υπόψη της το γεγονός ότι στη Νότια Ιταλία κλείνανε ε, βρεφονιπιακοί σταθμοί και ε, κέντρα για τους ε, υπερήλικες καπί και γυροκομεία. Άρα δηλαδή θα πρέπει κανείς να συνεχίσει να προσφέρει βασικές υπηρεσίες αυτές οι υπηρεσίες ας πούμε για τους ηλικιωμένους αυτές απαιτούν και ρυθμίσεις υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτές ακριβώς τις ημέρες λαμβάνουμε μέτρα που είναι αντικυκλικής μορφής όπως ε, οι παρεμβάσεις de minimis για τις μικρές επιχειρήσεις ή όπως οι παρεμβάσεις ε, για, ε, τους, για τα γραφεία ευρέσης εργασίας ή οι παρεμβάσεις όπου καταβάλλονται επιδόματα σε περιπτώσεις που τις χρειάζονται ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων. Τώρα, ε, τέτοιο το ερώτημα κατά πόσο είμαι ευχαριστημένος ή απογοτευμένος. Κοιτάξτε, ο υπουργό, ο υποφαινόμενος δηλαδή, είναι απογοτευμένος. Γιατί αν δείτε το γράφημα, ε, η εικόνα δεν είναι καλή, είναι πολύ επίπεδη. Άρα δηλαδή πρέπει να δεχτούμε ότι εντάξει ο στόχος του Μαΐου έγινε επιτεύχθηκε αλλά για να επιτύχουμε αυτό του Οκτωβρίου σε πολύ λίγες ημέρες πρέπει να επιτύχουμε άλματα. Αυτή όμως η δυναμική δείχνει ότι δεν υπάρχει καλή διαχείριση στην Ιταλία. Ε, πώς να είναι κανείς ευχαριστημένος αλλά αυτό είναι συνεπές με το ότι τουλάχιστον ε, ορίσαμε κάποιους στόχους. Άρα δηλαδή δεν είμαι ευχαριστημένο, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, διαπιστώνω ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε τους στόχους μας. Λίγο περίπλοκα, αλλά ε, συνδυασμένες αυτές οι δύο απόψεις που σας ανέφερα και ε, μέχρι τώρα έχουμε χάσει βέβαια, χάσαμε πέρυσι 1,5 εκατομμύριο. Τελευταία παρατήρηση για την Πομπία Για την Πομπία είπα ότι εμείς ε, προβλέπουμε να ανοίξουν ε, τα πέντε πρώτα εργοτάξια, όπως αποκαλούνται στην Ιταλία, ε, έτσι, αυτό θα γίνει το Δεκέμβρη μάλιστα, έτσι ώστε τον Ιανουάριο ελπίζω να ανοίξουμε την Πομπία. Αυτά τα, τα εργοτάξια θα χρηματοδοτηθούν από κοινωτικά προγράμματα. Γιατί όλα αυτά ήταν χρονοβόρα πάρα πολύ απλά, διότι η Πομπία βρίσκεται σε μία περιοχή του Νότου όπου υπάρχει πυκνότατη και διάχυτη εγκληματικότητα. Άρα δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε. Έπρεπε να εξασφαλίσουμε ότι οι διαγωνισμοί που θα προκυρήσονταν ε, το αποτέλεσμα τους ε, να μην ε, κατακυρώνονταν σε λάθος μέρος να μην χανόταν το ένα ευρώ. Αυτό ήταν ο, χώρο, ο λόγος. Η Ιταλική κυβέρνηση στο τέλος αυτού του έτους θα καταθέσει ένα έγγραφο ε, πρόσκλησης σε διάλογο το οποίο ξεκινάει από το πρόγραμμα εργασίας. Και όπως μπορείτε να φανταστείτε και εδώ, όπως και σε όλες τις άλλες χώρες, θα προκύψει μια ανοιχτή και ουσιαστική αντιπαράθεση. Σας κατευχαριστούμε. Όπως είπαμε και στον κύριο Χατζηδάκη, και εσείς είστε μέλος του Συμβουλίου. Φαίνεται ότι είστε υπερορισμένων στοιχείων της θέσης μας. Ελπίζουμε λοιπόν και στο Συμβούλιο να τα πείτε αυτά. γιατί έτσι μόνο θα βρεθεί συμβιβασμός αποδεκτός από όλους. Σας ευχαριστώ λοιπόν ακόμη μία φορά και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Κάποτε θα ξανάρθετε ελπίζω για να μας πείτε ότι υπήρξε και ακόμα περισσότερη πυρόδος